Να κάνουμε μια δοκιμή. Θα μιλήσω γερμανικά. Μ' ακούτε σε όλες τις γλώσσες. Οι κυρίες και κύριοι από την Ισπανία μ' ακούνε, καταλαβαίνουν. Ο γερμανικά πρέπει να μιλήσω, λέει ο μιλητή. Ισπανικά, αγγλικά, τα ελληνικά ακούγονται παρακαλώ. Σας καλωσορίζω και πάλι. Καλωσορίζω την ε, Ισπανίδα Υπουργό. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, να της δώσουμε το λόγο να μας ε, κάνει την ομιλία της ε, και κατόπιν θα θέσουμε ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ως Υπουργός Επιστημών και Καινοτομίας έχετε το λόγο και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το πρωινό μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας. Είναι τιμή μου και ικανοποίηση μου να είμαι ενώπιόν σα και να μπορέσω να σα εκθέσω ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητε που ε, έχουμε θέσει κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμεινο του 2010 από τη σκοπιά του Δικού μου Υπουργείου. Η δική μα Προεδρία συμπίπτει με ένα νέο σημαντικό στάδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη θέση ισχύ τη Συνθήκη Λισαβόνα την 1η Δεκεμβρίου και ε, ταυτόχρονα εμείς θα παραβρεθούμε και στη σύσταση της Νέας Επιτροπής ε, φέτος. Ε, κλείνει επιπρόσθετα ένας κύκλος που ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2000 με τη θέση ισχύ της στρατηγικής της Λισαβόνας, μια δεσμεύση των κρατών μελών για να καταστήσουν την Ευρώπη το 2010 την οικονομία που θα βασιζόταν στη γνώση, την πιο δυναμική και ανταγωνιστική του κόσμου, σεβόμενη την κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον δέκα χρόνια μετά και παρά το ότι η Ευρώπη συνεχίζει να έχει εκκρεμείς προκλήσεις, η στρατηγική μας επέτρεπε να συνενέσουμε σε ένα πολιτικό όραμα, να χαράξουμε πορεία και να θέσουμε κοινά θεμέλια ε, για την πρόοδό μα. Τώρα ανοίγουμε ένα νέο στάδιο που ε, θα χαρακτηριστεί από τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, μια στρατηγική που γεννιέται στο πλαίσιο μια ε, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο το πιο βαθύ πολιτικό προβληματισμό των τελευταίων δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να καταρτήσει ένα νέο οδικό χάρτη, ως πιο ρεαλιστικό από ό,τι στο παρελθόν, αλλά με έναν ε, στόχο ε, που έχει ήδη τεθεί στα πλαίσια στρατηγική Αβώνας, ε, την οριστική ανάπτυξη της κοινωνίας και οικονομίας της γνώση Είναι τόσο σημαντική η πρόκληση που ο πρόεδρο Μπαρόσο στις ε, προσανατολισμού για την επόμενη Κομισιόν υπογράμμισε την αναγκαιότητα η Ευρώπη να στοιχηματίσει για μια ριζική μεταμόρφωση προ ε, μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση. Ακόμη δεν ε, έχει αναλάβει καθηκοντά τη η νέα Κομισιόν, αλλά γνωρίζουμε πω θα δυναμηθούν οι αρμοδιότητε των τριγών τη γνώση στο Σώμα των Επιτρόπων, η δημιουργία ενό χαρτοφυλακίου που για πρώτη φορά αναλαμβάνει αρμοδιότητε τη επιστημών και σε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Υπουργείου μα μας μας δίνει ένα μήνυμα ολοκλήρωσης με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Μιλάμε για ένα θέμα πραγματικά στρατηγικό για την Ευρώπη, δίχως περισσότερες επιστήμες και καινοτομία και κυρίως δίχως ε, την απαραίτητη ολοκλήρωση και μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων η Ευρώπη δεν θα μπορέσει ε, να διατηρήσει την ηγετική της θέση ούτε να βελτιώσει ε, τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Προ την κατεύθυνση αυτή πιστεύω ότι τα δεδομένα τη μελέτη «Ο κόσμο το 2025» που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο μας δείχνουν πολλά. Ε, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, το 61% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι στην Ασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει μόνο το 6,5% του πληθυσμού. Η τριάδα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία θα χάσει την ηγετική τη θέση στο εμπόριο και την παγκόσμια παραγωγή και η Κίνα. Ε, σας είπα μόλις ότι έγινε η δεύτερη οικονομία ε, του κόσμου ε, μπροστά από την Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας δείχνουν ότι αν ε, δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα το 2025 οι περισσότερες επιστήμες ε, ε, θα ε, παράγονται εκτός από τις χώρες που μέχρι τώρα θεωρούνταν ε, ηγέτες και θα ξεπεραστούμε από την Ασία μόνο δύο χώρες η Κίνα και η Ινδία θα εκπροσωπούν το 20% της παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης δηλαδή το διπλό από το σημερινό ποσοστό τους στο πλαίσιο αυτό που είναι το πιο πιθανό να συμβεί σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία η Ευρώπη θα μπορέσει να διασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ε, διεθνή σκηνή αν δράσει στον τομέα επιστημών και καινοτομία με πιο ενωμένο και στιασμένο τρόπο στι προκλήσει. Το να πετύχουμε αυτήν την ενότητα δράση, αναμφισβήτητα αποτελεί πρόκληση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει από τι επαρχέ τη εμπόδια που φαίνονταν υπέρβλητα. Ε, καταστήσαμε πραγματικότητα τέσσερι πολύ σημαντικέ ελευθερίε, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ατόμων και κεφαλαίου σε μια Ευρώπη σχεδόν 500 εκατομμυρίων κατοίκων με 27 χώρε και ένα νέο νόμισμα για 16 από τι χώρε, αυτέ που χρησιμοποιείται πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα. Είναι η στιγμή να προχωρήσουμε σε μια νέα διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενότητα που ήδη είναι γνωστή ω η πέμπτη ελευθερία ή η ελευθερία Κυκλοφορία τη γνώση και του ταλέντου γιατί μόνο σε ένα κοινό χώρο για τη γνώση, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ε, όπου οι επιστήμονες και οι ιδέες θα κυκλοφορούν ελεύθερα, μπορούμε να εγγυηθούμε αυτή την κοινωνία και αυτή την οικονομία της γνώσης που επιθυμούμε για την Ευρώπη. Η Ισπανία μαζί με τις χώρες ε, του Τρίτου Προεδριών, Βέλγιο, Ουγγαρία, παίρνει τη σκητάλη από τη Σουηδία και τις προηγούμενες προεδρίες, συνεχίζοντας με ενθουσιασμό και φιλοδοξία τα καθήκοντα αυτά. Οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας ό,τι αφορά την έρευνα διαρθρώνονται ε, στο να προωθήσουμε αυτό αυτές τρει διαστάσει διαστάσεις του ευρωπαϊκού χώρου έρευνα, δηλαδή την ολοκλήρωση, την εμπλοκή και την ένταξη όταν ε, μιλάμε για την ολοκλήρωση αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα να θέσουμε τις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας ε, στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Πρέπει να πετύχουμε ε, ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να λειτουργήσει ως ενέος χώρος και θα έχει, να έχει δεσμικό βάρος, να μην υπάρχουν νέες γραφειοκρατικές δομές, αλλά μηχανισμοί που θα μας βοηθήσουν να ε, αποφύγουμε τις ε, διπλές προσπάθειες ε, και να ευθυγραμμίσουμε τις προτεραιότητες των κρατών μελών. Θέλουμε να βελτιώσουμε την διαχείριση αλλά και να προωθήσουμε τις πέντε πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των ερευνών και να διευκολύνουμε την κινητικότητά τους. Επίσης θα προωθήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο έρευνας μέσα από υπηρετικές συνδιασκέψεις που θα επιτρέψουν να προωθήσουμε την προοπτική όλων των πρωταγωνιστών στον του τριγώνου της γνώσης. Επίσης, ε, θα σημειώσουμε πρόοδο σε συγκεκριμένες πτυχές ε, ε, που θα καταστήσουν ερωτώ αυτό τον ενιαίο χώρο αυτή της πέμπτης ελευθερίας με προτάσεις για να εξελίψουμε τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα για την κινητικότητα ή θα αναπτύξουμε ένα δίκτυο υποδομών επιστημονικών και θα αναπτύξουμε το χάρτη ΕΣΦΡΕ, Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρο Ερευνητικών Υποδομών ή θα προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Αλλά η δική Είμαστε μας διάσταση για την ολοκλήρωση υπερβαίνει τα σύνορα και αναζητά συνεργίες και υφιστάμενες συνδέσεις μεταξύ αυτής και των ε, τομέων του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καινοτομία. Θέλουμε οι συζητήσεις ε, και για τα δύο ζητήματα να αλληλεπιδράσουν ε, μεταξύ, να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικού και βιομηχανικού τομέα και φυσικά οι υπουργοί στην διασκέψη θα χρησιμεύσουν τα μάλα γι' αυτό. Ε, ήδη το πράττει η Ισπανία βέβαια μέσα από το Υπουργείο του οποίου είμαι υπεύθυνη. Ε, η, στρατη... η Ισπανία αυτή τη στιγμή εργάζεται ήδη για νέα μια στρατηγική καινοτομία ε, που προσεγγίζει σαφώ τη σχέση μεταξύ καινοτομία και επιστήμη και ε, θέτει πέντε άξονε προτεραιότητα. Ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον ευνοϊκό για την καινοτομία, τι lead market για τι δημοσίε αγορέ ω ατμομηχανέ για την καινοτομία, διεθνοποίηση τη καινοτομία, διάδοση τη καινοτομία ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τέλος ε, τα άτομα ως ε, άξονας του, της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Από την άλλη θέλουμε να συνεισφέρουμε στην παγίωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνα στο ET, στηρίζοντας την λειτουργία των πρώτων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομία, των ΚΙΚΣ, οι οποίες, έχουν, οι οποίες θα συνεργάζονται με, για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας ε, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά μόνο αν θεωρήσουμε ότι ο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα είναι ακρογωνίο λίθο για τη μελλοντική στρατηγική 2020. Προτείνουμε στρατηγική για το 2020 να συμπεριλαμβάνει δείκτε και στόχου από τη σκοπιά του αέρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να εκφράζουν το όραμα τη Λισαβόνα για να εντάξουν πέρα από τι επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη και ε, αξιολογήσει των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των επενδύσεων αφού περιέγραψα τον άξονα της ολοκληρωσής που είναι ο πιο πληρής, ε, θα περάσουμε στο δεύτερο άξονα ε, την εμπλοκή με δύο λόγια. Ε, θέλουμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, να, να παρουσιάσουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επιστήμη στις καθημερινές μας ανησυχίες, στις προκλήσεις και στην ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη. Ε, στο άτυπο συμβούλιο θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε μια κοινή θέση για το θέμα αυτό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιστήμης και κοινοτομία θα πρέπει να εμπλακούν ε, ε, πιο αποφασιστικά στο να απαντήσουν τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι νέες πηγές ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, επίση επί των φυσικών πόρων, η γύρανση του πληθυσμού και οι σχετικές νόσοι, η αυξανόμενη διεθνής ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης δεν μπορούμε να περιμένουμε να παγιώσουμε τον αέρα για να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι έχουμε επαρκή εργαλεία σήμερα για να προχωρήσουμε και πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά του Ω συγκεκριμένη πρωτοβουλία θέλουμε να προωθήσουμε την απλούστευση τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο έτσι ώστε το διοικητικό άχθο ε, να μην ε, αποτελεί ε, ουσιαστικά κόλλημα για τις ομάδες έρευνας και τις επιχειρήσεις. Ε, ουσιαστικά σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, δραστηριότητες αυτές οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις αποτελούν την κυρία πηγή απασχόληση στην Ευρώπη και μέσω αυτών θα οικονομήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που να βασίζεται περισσότερο στη γνώση. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στη στήριξη και παγίωση των νέων επιχειρήσεων με τεχνολογική βάση όπως και αυτών των ΜΜΕ που θέλουν ε, να επαναφευρεθούν χάρη στην καινοτομία σε παραδοσιακού τομεί. Επίση, προτείνουμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα Έρευνα να προωθήσουμε πρωτοβουλίε που να απαντούν στο πνεύμα αυτό εμπλοκή, όπω ε, είναι η περίπτωση των ε, συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του ε, σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, ε, το πράσινο αυτοκίνητο, το διαδίκτυο του μέλλοντος, τα εργοστάσια του μέλλοντος, και ε, κατασκευές. Θα ήθελα τέλο να επισημάνω ότι η Ισπανική Προεδρία εργάζεται σε δύο, επί δύο νομοθετικών προτάσεων για το GMS και το bonus, ε, όπου έχουμε συναπόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για να κλείσω με την περιγραφή του πρωτοτήτου η τρίτη διάσταση του ΕΡΑ, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα ε, είναι η ένταξη ένα σημαντικό αριθμό ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, και η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας ε, βιώνουν, μια, βιώνουν σημαντικές ελλείψεις και θεωρώ ότι μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο εγγύς μέλλον μέσα από την επιστήμη και την καινοτομία. Θέλουμε να υπερασπίσουμε ότι η Ευρώπη της γνώσης πρέπει να εργαστεί για μια επιστήμη με μεγαλύτερη ευαισθησία που μεταξύ των προκλήσεων θα συμπεριλαμβάνει την παγκόσμια διάδοση τη επιστημονική γνώση με συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που θα απευθύνονται σε ομάδε και χώρε με μεγαλύτερε δυσκολίε για την πρόσβαση στη γνώση αυτή, το κοινωνικό αντίκτυπο ε, και την εστίαση στην ανάπτυξη τη αξιολόγηση τη σχεδίαση και του σχεδιασμού. Μια επιστήμη η οποία θα θέλει να διαβάσει τεχνολογία στι ε, ε, πιο ευάλωτες ε, περιοχές του κόσμου ε, και ε, αναφέρομαι στην καταπολέμηση επίσης του ψηφιακού κάσματος και στην παγκόσμια πρόσβαση σε φάρμακα και τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Έχουμε οργανώσει για όλα αυτά μια διεθνή συνδιάσκεψη για την επιστήμη κατά της φτώχειας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο και ελπίζουμε ένα μέρος των συμπερασμάτων να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Συμβούλιο Διαγωνιστικότητας του Μαΐου. Ένας άλλος τρόπος ε, να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Ε, πέρα από το ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια Συγγνώμη, περισσότεροι πανεπιστημιακοί και διδακτορικοί είναι γυναίκε. Αυτέ μόνο καλύπτουν το 17% των θέσεων υψηλή ευθύνη θα πρέπει η εστίαση στο φύλλο να ενταχθεί στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των πολιτικών επιστημών. Κυρίες ε, και κύριοι, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, γνωρίζουμε το πρόγραμμά μας ε, ουσιαστικά περιορίζεται χρονικά, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας για να το ολοκληρώσουμε. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας για την ολοκλήρωση, την εμπλοκή και την ένταξη, ελπίζουμε να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ συγκεκριμένες πτυχές που έχουν να κάνουν με την βασική έρευνα αριστείας, τις ευκαιρίες ευκαιρίες ε, για ε, τους ε, ερευνητές, τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Επιστημονικών Υποδομών, την σύνδεση των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και την χορήγηση ευκαιριών των αποκλεισμένων έτσι ώστε η καινοτομία και η ανάπτυξη να απαντήσει στις ανάγκες τους. Η δική σας συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες αυτές τις προκλήσεις είναι απαραίτητη και η Ισπανία θα ήθελε να ευχαριστήσει εκ των προτέρων ε, να σας ευχαριστήσω και προτείνω για τη δέσμευσή σας και τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας και θα δράξουμε την ευκαιρία τώρα να θέσουμε ερωτήσεις. Ήδη έχουμε μακρύ κατάλογο ανθρώπων που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Προτείνω λοιπόν ε, να περιοριστούμε σε ένα-δύο λεπτά, ώστε όλοι να έχουμε ε, την ευκαιρία να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Ε, η κυρία Καστίγιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους της ομάδας μου, καλώς ήλθατε στην Επιτροπή αυτή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστούμε για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και για την παρουσίαση των στόχων της Ισπανικής Προεδρίας ό,τι αφορά την ε, έρευνα και την καινοτομία. Γνωρίζουμε όλοι το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η έρευνα και καινοτομία στο μέλλον ε, της κοινωνίας και μάλιστα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αλλά πέρα από όλες τις δυσκολίες ε, της ε, ανάπτυξης της έρευνας, ένα από τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε και που συστηματικά προκύπτει ανά διάφορες περιόδους και στην ίδια την περίοδο του προγράμματος πλαίσιο είναι η πολυπλοκότητα των κανόνων που πρέπει να γίνουν σεβαστοί για να μπορέσει κάποιο να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό ισχύει και για του ερευνητέ αλλά και για τι ΜΜΕ θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει μόνο μία απογοήτευση, γιατί πάντοτε υπάρχει μία υπόσχεση για ουσιαστική βελτίωση και τι συμβαίνει τελικά. Δεν ε, λαμβάνει χώρα αυτή η βελτίωση. Θεωρείται θετικό αυτό που συνέβη ε, στη μετάβαση από το έκτο στο έβδομο πρόγραμμα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες. Δεν μπορεί η έρευνα ε, να πρέπει να περάσει από μία οδό για τα κολλήματα, όταν μπορούν να έρθουν ε, αυτά τα κολλήματα σχετικά εύκολα πιστεύω εγώ. ένα πραγματικά με αγγίζει η προσέγγισή σας για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, η ευαισθησία σας. Μπορείτε να μα εξηγήσετε συγκεκριμένα ποια μέτρα σκέφτεται να υλοποιήσει η Ισπανική Προεδρία για να υπερβληθούν κάποιε από αυτές τις θεμελιώσεις δυσκολίες. Danke, Frau Muchas Κυρία Μαδουρέλ, ευχαριστώ. Και εγώ, εξ ονόματο τη ομάδα μου, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σα καλωσορίσω στην Επιτροπή αυτή και να σα συγχαρώ για την παρουσίασή σα, που πιστεύω ότι καθιστά ε, σαφή τη δέσμευση τη Ισπανική Προεδρία στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σα θέσω κάποιε ερωτήσει ε, σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν αυτή την Επιτροπή και επί των οποίων πιστεύουμε ότι χρειάζονται νέε ιδέε, καινοτόμε ιδέε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Ουσιαστικά συνάδει αυτό με την ερώτηση τη συναδέλφη, δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ τη έρευνα και του παραγωγικού τομέα. Εσεί, ε, βάσει τη προσωπική σα διαδρομή, γνωρίζετε πολύ καλά τόσο τον ακαδημαϊκό κόσμο όπω και τον επιχειρηματικό. Ε, ήσασταν ε, ερευνήτρια και επιτυχής επιχειρηματίας ε, στον τομέα της βιοτεχνολογίας, πολύ σημαντικό τομέα. Και μπορείτε να συνεισφέρετε τα μάλα με την προσωπική σας εμπειρία όταν μιλάμε για ανάληψη πρωτοβουλειών, για την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Αυτό είναι θεμελιώδες και όλοι συμφωνούμε σε αυτό και το είπατε κι εσείς, για να ενδυναμώσουμε και την έρευνα όσο και την καινοτομία. Ε, ε, ουσιαστικά μας παρουσιάσετε τις ιδέες Ισπανικής Προεδρίας. Ε, αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, από τη δική, βάση της δικής σας εμπορίας, ποια μπορεί να είναι τι θα κάνει μάλλον η Ισπανική Προεδρία για να βελτιώσει το διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκού διαλόγου και επιχειρήσεων, κυρίως με τις ΜΜΕ Ίσως ε, αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πολύ σύντομα, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ε, μας ε, φαίνεται πολύ στοχευμένο αυτό η προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας να προωθήσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας δηλαδή, αλλά αυτό στην πράξη απαιτεί πολλά, ε, πρέπει να επιληθούν πολλά προβλήματα, το αναφέρατε κι εσείς, είπατε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά για εργασίας για τους ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο για τη σταδιοδρομία των ερευνητών και πρέπει να καταργηθούν και τα εμπόδια για την ε, κινητικότητα των ερευνητών, ε, είτε διατομεακά είτε γεωγραφικά εμπόδια. Πώς σκέφτεται η Ισπανική Προεδρία να προχωρήσει στο θέμα αυτό, κυρίως ε, ό,τι αφορά την εξάλληψη των κολλημάτων στην κινητικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Φιονκέρης. Ε, Καλημέρα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Και ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω εκ μέρους της ομάδας μου, της ομάδας των Πρασίνων. Και φυσικά χωρίς ε, να ε, είμαστε γενείς θα ήθελα καλά να σας υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο σας περιόρισε τον προϋπολογισμό για την έρευνα και νομίζω ότι κάποια στιγμή εσείς είπατε ότι όχι μόνο είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τον όγκο και το ποσοστό των επενδύσεων στην ε, έρευνα, αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι λοιπόν, προς αυτήν την κατεύθυνση από τη δική μας ομάδα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια κριτήρια μπορούμε να θεσπίσουμε για να μετρήσουμε αυτή την αποτελεσματικότητα της διαβίβασης της γνώσης. Και επίσης να ρωτήσουμε αν έχετε κάποια σχετική πρόταση. Και πολύ σύντομα και ταπεινά, επιτρέψτε μου μία πρόταση, όχι μόνο σε εσά, αλλά στο Συμβούλιο και ίσως σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δηλαδή, ίσως ένα μέσο για την προώθηση αυτής της διαβίβασης της γνώσης, για την απόπειρα αξιολόγηση αυτής της διαβίβασης της γνώσης, θα μπορούσε να είναι το εξή δεδομένου ότι σε πολλά κράτη οι ερευνητές είναι οι ε, καθηγητές στο πανεπιστήμιο, ή θα μπορούσε να γίνει αξιολόγηση τους ε, για τη διάδοση της ε, γνώσης. Σε κάποια κράτη γίνεται αυτή η αξιολόγηση, αλλά σε πολλά άλλα κράτη δεν ε, ε, υπάρχει αυτό το κούρσους όνουρ για την αξιολόγηση. Η Αγγέλικα Νίμπλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία, Πρόεδρε, σας ε, Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ε, ήρθατε. Δύο θέματα θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχήν μιλήσατε για ολοκλήρωση και συμμετοχή της ε, επιστημονικής κοινότητας. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν σε όλα τα προγράμματα που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα έρευνας του EIC, του EIT. Νομίζω ότι είναι πάντα σημαντικό να τονίζουμε ότι το μόνο κριτήριο σύμφωνα με το οποίο δίδονται τα πόροι για την έρευνα θα πρέπει να είναι το κριτήριο της αριστείας. Ε, και θα ήθελα να ρωτήσω εάν συμφωνείτε. Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ε, που έχει ξεκινήσει τις ε, εργασίες του επίσημα. Ε, παρακολουθείτε από, την, το Κοινοβούλιο μας και είμαι η συγγήτρια για το θέμα. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του Ιουνίου πέρσι υπάρχει και βλέπω στην έκθεση αυτή ότι η, πρόκειται για ιστορία επιτυχίας. Ήδη στους ε, διαγωνισμούς είχαμε ε, πολλούς υποψηφίους. Ε, Πρόκειται λοιπόν για πολύ θετική ιστορία και Πιστεύω ότι έχει αποδείξει την αξία του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει πληθώρα ελλείψεων, ε, διαχειριστικών ελλείψεων και η πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι μια μακροπρόθεσμη τροποποίηση της δομής αλλά και βραχυπρόθεσμα να ε, παράσχουμε οργανωτική βοήθεια. Υπάρχει μια μακρά σειρά ε, συστάσεων και ε, θα σας ε, ε, όπου μας παρακαλούν να γίνουν γρήγορα αλλαγές και η ερώτησή μου είναι τι θα κάνετε εσείς βραχυπρόθεσμα, τι θα γίνει για να γίνει πιο επιτυχής η δουλειά του ERC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Τσουκάλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό στην αρχή της, Ευρωπαϊκής της Ισπανικής Προεδρίας να ακούσουμε ποιες είναι οι απόψεις σας. Κατάλαβα από τους αριθμούς που θέσατε ότι έχετε υπόψη σας την μελέτη Global Trends in 2025 εκεί όπου περιγράφεται η αποτυχία του κλασικού, των κλασικών ηγετικών δυνάμεων της έρευνας του σήμερα να συναγωνιστούν τις χώρες BRIC το 2025. Όμως αναφέρατε και μερικά πολύ σημαντικά ζητήματα. Αναφέρατε το γεγονός ότι η Ευρώπη ε, έχει ένα πολυπίκυλο ερευνητικό τοπίο και ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε μια κοινούς άξονες με τους οποίους να επιχειρήσουμε την ερευνητική μας προσπάθεια. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε σχέση τόσο με την καινοτομία όσο και με την πολιτική έρευνας ε, δεν είναι απλώς πολυπίκυλο, είναι περίπου σουρεαλιστικό. Έχουμε 29 δράσεις, 9 προτεραιότητες, 2 πολιτικές και συνεπώς υπάρχει εκτός από αυτό που αναφέρει η κυρία Νίμπλερ η πολυπλοκότητα ε, και η κυρία Πιλάρ Δεκαστήγιο η πολυπλοκότητα για τη χρηματοδότηση ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαστε επικεντρωμένοι στις διαδικασίες και όχι στον έλεγχο, στην αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Θα ήθελα να σας πω ότι η Σουηδική Προεδρία εξέδωσε ε, ένα κείμενο το οποίο λέγεται A European Paradise, στο οποίο ασκεί κριτική για τα τις κύριες παθογένειες του ελληνικού ερευνητικού του ε, ευρωπαϊκού συστήματος. Εκεί λέει ότι 2.000 ε, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δίνουν διδακτορικά, 180 δίνουν στην Αμερική και 120 στην Κίνα. Και τέλος λέει ότι καλό θα είναι αντί για αγροτικές επιδοτήσεις, που είναι η κύρια ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασχοληθούμε με τις επιδοτήσεις της έρευνας και η ερώτηση μου είναι προς την ενοποίηση του πολυσχηδούς και πολυειδούς αυτού ε, ερευνητικού τοπίου. Πώς θα εργαστεί η Ισπανική ε, Προεδρία για να επιφέρει μια ομογενοποίηση για να στις προθέσεις της είναι η αριστεία και η επιλεκτικότητα στις χρηματοδοτήσεις, ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών θα αποτελέσουν έναντι της συνοχής μια υπέρτερη επιλογή. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καβάλιο. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Μία ναι, από τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρώπη είναι η δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Αναφερθήκατε στην κινητικότητα και στις μεγάλες υποδομές. Εγώ θα ήθελα να ε, προσθέσω και το κοινό πρόγραμμα. Ε, είχαμε μέχρι σήμερα εμπειρίε από το ΕΡΑΝΕΤ και το άρθρο 169. Υπάρχουν όμως προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μεγάλο γραφειοκρατικό άχθο και με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Πώς βλέπετε τη μελλοντική ανάπτυξη αυτών των κοινών προγραμμάτων κρατών μελών και επιτροπής, ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας ή το, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Στούτο Τεχνολογίας ε, θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε μετα πανευρωπαϊκά προγράμματα με ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση. Ε, ουσιαστικά ε, η χρήση των ε, μέσων αυτών στην οικοδόμηση και παγίωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου θα είχε πλεονεκτήματα. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Υπουργέ να τοποθετηθείτε για αυτές τις δυνατότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα την ευκαιρία στην Υπουργό να απαντήσει στις ερωτήσεις του πρώτου τμήματος και κατόπιν θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ομαδοποιήσω τις ε, παρεμβάσεις. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας και για τις προτάσεις σας. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, νομίζω ότι αν μπορέσει η Ισπανική Προεδρία να συμβαδίσει με την Κομισιόν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της απλούστευσης, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα στην Ευρώπη. Άλλωστε πρόκειται για ένα προβληματισμό που πρέπει να γίνει από κοινού με όλα τα όργανα και με το ελεκτικό συνέδριο. Θα αναμένουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις, δεσμευτικές αποφάσεις, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει ε, σε έναν προβληματισμό που να έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις επιχειρήσεις μας και τους ερευνητές μας ε, και αυτό μπορεί να γίνει αν είμαστε λιγότερο γραφειοκράτες από την αρχή και με φυσικά με μια ισχυρότερη αξιολόγηση και έλεγχο στο τέλος, έτσι ώστε να ε, καθιστούμε υποχρεωτική την ολοκλήρωση ε, των ε, σχεδίων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε καταρχήν πού μπορούμε να εξελίψουμε τη γραφειοκρατία. Και δεύτερον, να προχωρήσουμε στην εστίαση των ε, μέσων. Εγώ νομίζω όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν ε, θέσει σε εφαρμογή νέα μέσα και νέα προγράμματα. Όλοι ξέρουν ε, πόσο συναρπαστικό είναι να ξεκινά κανείς ένα νέο πρόγραμμα αλλά τελικά μερικές φορές πρέπει να λέμε ότι αυτή η προσκλήση υποβολής προτάσεων τελικά πρέπει να κλείσει, μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει όλα τα διαφορετικά μέσα που έχουμε ε, και μπορούν να μας εξυπηρετήσουν ε, στην επίτευξη των στόχων μας. Είναι η Ευρώπη προχωρήσει προς λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα προγράμματα, αλλά εστιάσει περισσότερο στους στόχους, νομίζω ότι θα κάνει ένα μεγάλο βήμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είναι ένα θέμα που το γνωρίζω καλά γιατί πέρα από το ότι προέρχομαι από το τομέα της ε, βασικής έρευνας ε, ήμουν και επιχειρηματίας σε μια ομάδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Έτσι λοιπόν ε, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να έχει κανείς πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το να μπορούμε να ε, απλοποιήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες θα είναι ένα μεγάλο βήμα λοιπόν ε, και να μπορέσουμε να έχουμε ε, ισχυρές, μεγάλες πρωτοβουλίε στον τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι οποίε θα συμμετέχουν και μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Γι' αυτό, στον άξονα της Προεδρία που αφορά την εμπλοκή, implication, προωθώντας ε, τον κοινό προγραμματισμό και τις ΔΙΤ. Εκεί έχουμε δύο άξονες όπου οι ΜΜΕ μπορούν να διδραματίσουν ένα πολύ σχετικό σκόπιμο ρόλο. Δηλαδή θέλουμε οι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει να εστιάσουν τι μεγάλε προκλήσεις που έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε και να μπορέσουν ε, να προσανατολιστούν ε, σε ό,τι φορά τη διαβίβαση της γνώσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο έρευνα. Καταρχήν, Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να εξελίψουμε τα παραδοσιακά μοντέλα. Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας που είναι μεγάλη πρόκληση, μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να θέσει τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένες ε, αρμοδιότητες ε, που δεν ε, εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο των Υπουργών Επιστημών. Εμείς θα δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να βελτιώσουμε τη στεδιοδρομία των ερευνητών και την κινητικότητα. Πρέπει να εργαστούμε συγκεκριμένα για την πρόθεση αυτής της πέμπτης ελευθερίας στο Συμβούλιο του Μαΐου οι Υπουργοί Επιστημών θα πρέπει να μπορέσουμε να παρέμβουμε και σε συμβούλια, άλλα υπουργικά συμβούλια ε, όπου υπάρχουν ε, αρμοδιότητες ε, που να αφορούν τον τομέα των επιστημών. Θα υπάρχει ευκαιρία να τεθούν αυτά τα ε, θέματα στο Συμβούλιο Απασχόληση, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Νομίζω ότι πρέπει οι Υπουργοί να καταλάβουν ότι θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στο Σώμα των Ερευνητών ε, ε, που πρέπει να χαίρουν υψηλή κινητικότητα ε, και για να υπάρχει αυτή η κινητικότητα πρέπει να αρθούν τα κολλήματα στην κινητικότητα των ερευνητών. Ε, θα εξετάσουμε το πώ οι ερευνητέ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε στα διάφορα συστήματα ε, κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση που υπάρχουν σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και να δούμε πώ θα εγγυηθούμε ότι πώ αυτή η κινητικότητα η κινητικότητα μάλιστα είναι υποχρέωση ε, των ερευνητών, αλλά είναι και δικαίωμά τους. Α δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη, βελτι... τη των ερευνητών, γιατί κάτι τέτοιο το χρειάζεται η Ευρώπη για την ανταγωνιστικότητά της. Τώρα, βάσει της δικής μου πείρας, για <laughs> τη σχέση που υπάρχει μεταξύ καινοτομία και επιστήμης. Νομίζω ότι εδώ και δύο χρόνια μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και σχετική εμπειρία στο Υπουργείο. Πρώτη φορά η Ισπανία θέτει στο δύο χαρτοφυλάκιο καινοτομία και επιστήμες και μπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Μία πρώτη δράση είναι ο κοινό προβληματισμό, ο κοινό στοχασμό. Και νομίζω ότι με τον έρευνα, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα, προχωρήσαμε πολύ και νομίζω ότι αυτή η πρόοδος θα πρέπει να αντικατοπτριστεί ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καινοτομία. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα κοινό στοχασμό και ακαδημαϊκοί αλλά και επιχειρηματίες θα πρέπει από κοινού να σκεφτούν για τους ίδιους στόχους. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες γέφυρες μεταξύ του κόσμου των επιστημών και της καινοτομίας Βέβαια, δεν πρέπει όλη η επιστήμη να επικεντρώνεται στην έρευνα, ούτε στην καινοτομία, με συγχωρείτε, ούτε όλη η καινοτομία πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη. Όμως υπάρχουν κάποια σύνολα και πρέπει να μελετήσουμε πώς μέσα από αυτά μπορούμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Το θέμα της κινητικότητας λόγου χάρη των ερευνητών, για το οποίο εργαζόμαστε ήδη στην Ευρώπη θα πρέπει ε, να το προωθήσουμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα κράτη-μέλη. Κινητικότητα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα λόγου χάρη και πρέπει να υπάρχει και κινητικότητα μέσα στο δημόσιο τομέα. Ε, τα επιστημονικά μεταξύ επιστημονικών Ινστιτούτων και πανεπιστημίων λόγου χάρη. Αυτό είναι κάτι επί του οποίου εργαζόμαστε στην Ισπανία και νομίζουμε ότι και στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχει διασφάλιση τη κινητικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τώρα και τα μέσα για τη χρηματοδότηση τη επιστημονική επιστήμης και της Αν δούμε, υπάρχουν ε, κάποια διαφορετικά μέσα, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός της αξίας της γνώσης από τη στιγμή που παράγεται μέχρι να μεταφραστεί σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και αυτός ο κοινό σχεδιασμός με διαφορετικά μέσα, αλλά που το ένα να βασίζεται στο άλλο, είναι ένας στοχασμός που θα μας βοηθήσει να παγιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Σε σχέση τώρα με την παρέμβαση του κύριου Χορκέρα, για το θέμα της μέτρησης. Νομίζω ότι πρέπει να σημειώσει πρόοδο η Ευρώπη. Όλα τα κρατημέλη μελη ε, ζουν την αναγκαιότητα, υπάρχει, μάλλον όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί αυτό το 3%. Και φυσικά αυτό βοήθησε στα ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύουν ένα τμήμα του προπολογισμού σε δραστηριότητε καινοτομία και έρευνα. Δεν κατορθώσαμε να εμπλέξουμε με τον ίδιο τρόπο και τον ιδιωτικό τομέα, έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί το 2000, αλλά σημειώσαμε πρόοδο. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να δεσμευτούμε στο να αποδείξουμε ότι οι επενδύσεις αυτές είναι αποδοτικές. Και αυτό από την κοινωνική, και, αλλά και από την οικονομική σκοπιά. Και έτσι λοιπόν ε, πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες παραμέτρους που να έχουν να κάνουν με την πρόοδο της, ε, των επενδύσεων, γιατί αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να σκεφτούν όχι ότι πρέπει μόνο να ξοδέψουν, αλλά πρέπει να ξοδέψουν καλύτερα και πολλά πρέπει να γίνουν βέβαια σε ό,τι αφορά το θέμα της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πρέπει να ξοδεύουν καλύτερα και επίσης πρέπει να απαντήσουμε στους πολίτες μας γιατί και για ποιο λόγο. Ποιοι είναι οι στόχοι των επενδύσεων αυτών, ποια είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις επενδύσεις αυτές. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε ορατό. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με τη διάδοση της επιστήμης, του πολιτισμού. Και νομίζω ότι τόσο στον τομέα της διάδοσης αλλά και στον τομέα ε, των δραστηριοτήτων της συνεργασίας για την ανάπτυξη αυτό πρέπει να αντεκοτρίζεται ε, και στα προγράμματα των ερευνητών. Οι επιστήμονες θα πρέπει να εμπλέκονται ε, στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει να δείχνουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ανταγωνιστικότητας ε, του ερευνητικού τομέα. Αυτή η συζήτηση που είχαμε για τα διάφορα μέσα από την αριστεία και τη συνοχή. Θα αναφερθώ και ε, στο ρόλο του ΙΑΣΥ. E η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική αν ε, δεν υπάρχει ταυτόχρονη πρόοδος στην αριστεία και στη συνοχή. Δεν ε, θα υπάρχει πρόοδος αν δεν υπάρχει συνοχή στην Ευρώπη, όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι στους δύο τομείς έχουμε διαφορετικά μέσα για να προχωρήσουμε. Η σύσταση της ε, ERC είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα που δείχνει ε, πώς η Ευρώπη δημιουργεί ένα μέσο που έχει να κάνει με την αριστεία. Είναι μεγάλη πρωτοβουλία αυτή και νομίζω ότι η Ισπανία έχει δεσμευτεί πλήρως ε, θα βοηθήσει να εφαρμοστούν οι συστάσεις ε, του ε, γνωμοδοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ίδια τη δομή αλλά και την απλούστευση. Και στις συζητήσεις ε, που έχουμε νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Πιστεύουμε ότι το ERC αποτελεί κλειδί για να προωθήσουμε ε, την αριστεία της Ευρώπης στον ερευνητικό τομέα. Αλλά έχουμε και την πτυχή της συνοχής και έχουμε και άλλα μέσα. Έχουμε στην Ισπανία τη συνοχή των περιφερειών μας. Ε, χρησιμοποιούνται ε, τα διαφορετικά ταμεία. Έχουμε πολύ σαφείς δείκτες πως μέσα από τις επενδύσεις των ε, κονδυλίων αυτών οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές μπόρεσαν να ε, προχωρήσουν, να σημειώσουν πρόοδο στο θέμα της βελτίωσης των υποδομών και προς την αριστεία. Γιατί πρέπει να δώσουμε κίνητρα ε, οι περιφέρειες αυτές που μπορούν να λάβουν κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής να θέσουν στόχους προς την αριστεία και να προχωρήσουν προς την αριστεία μέσα από εργαλεία συνοχής. Κατόπιν για το θέμα του κοινού προγραμματισμού. και για τις ε, συμπράξεις ιδιωτικού τομέα, PPPs. Ε, εδώ επισέρχεται ο άξονας της εμπλοκής, implication σε μια οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Και εγώ νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη αυτή η οικονομική συγκυρία. Η Ισπανική Προεδρία πρέπει να έχει συγκεκριμένη προσέγγιση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η στιγμή να καταστήσουμε όρατο ότι η επιστήμη μπορεί να επιφέρει λύσεις μέσω πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα. Ε, πολλά έτη ε, επενδύει η Ευρώπη στην ε, έρευνα και στην ανάπτυξη και μπορούμε τώρα να δείξουμε ότι έχουμε λύσεις τώρα να παρουσιάσουμε για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε ορατό με μια δήλωση του Άτυπου Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου στο Σαν Σεμπαστιάν, μια δήλωση που θα έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή, να θέσουμε ουσιαστικά την επιστήμη ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να έχουμε μία πιο αποτελεσματική επιστήμη η οποία θα απαντά στις παγκόσμιες προκλήσεις. Πρέπει να προωθήσουμε τα ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και πρέπει να παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή της Προεδρίας ε, που θα το λέμε Science for Recovery, δηλαδή επιστήμη για την ανάκαμψη εδώ και τώρα. Θέλουμε να διανεμηθεί η πρόταση αυτή και στους ε, Υπουργούς Βιομηχανίας, έτσι ώστε να δείξουμε στους Υπουργούς Βιομηχανίας ότι η επιστήμη θέλει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση όλων αυτών μεγάλων προκλήσεων που βιώνει τώρα η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Πρόβλημα χρόνου έχουμε τώρα. Θα μπορέσουμε μόνο να προλάβουμε εάν ο καθένας περιοριστεί στο ένα λεπτό. Όποιος έχει να κάνει ερώτηση, παρακαλώ να περιοριστεί στο ένα λεπτό. Η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χάρηκα για την πεποίθηση που εκφράζετε στις δηλώσεις σας. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. καθώς έχουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης της κινητικότητας, γιατί μεταξύ άλλων οι ερευνητές έχουν τη συνδρομία τους, θεωρούν ίσως ότι δεν χρειάζεται να κινηθούν. Δεύτερο, πολλές φορές τα πανεπιστήμια δεν κάνουν τίποτα με την κινητικότητα αυτή και αυτό για πολλούς λόγους. Δεν θα ήταν δυνατό στον ε, ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και στα κοινά προγράμματα να δημιουργηθούν κάποια μάστερ που να συνδέονται με διεθνή προγράμματα έρευνας, με υποτροφίες για διδακτορικά ε, και έτσι ώστε να είναι πλήρες ε, ε, αυτό το σύστημα κατάρτισης, ε, δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποια μάστερ και από πίσω ίσως να κρύβεται και κάποια επιχείρηση αν είναι απαραίτητο και φυσικά να δίνονται και υποτροφίες. Ε, Köszönöm, elnök úr. a Itt vagyok. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ και χαίρομαι για την παρουσίασή σας που ακούσαμε. Μου άρεσαν πολύ αυτά που άκουσα. Στην Ισπανία νομίζω ότι το Υπουργείο σας βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Μία ερώτηση έχω. Τι άποψη έχετε για το εξής. Στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, διατίθενται πολύ διαφορετικά ποσά για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην Σλοβακία μόλις 2% του ΑΕΠ, σε άλλα κράτη-μέλη 3 με 4%. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τις ε, διαφορές αυτές που υπάρχουν, να εξαλείψουμε τις ε, διαφορές και να πετύχουμε ισορροπία. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά η Ισπανική Προεδρία. Ερωτήσεις έχω όσον αφορά την, ε, την ε, συνοχή και την αριστεία. Από τις κάτω χώρες προέρχομαι Ε, Νίστερ Ρόι λέγομαι. Ε, εν πάση πτώση, μιλήσατε λοιπόν για αριστεία και για συνοχή. Ε, ποιοι θα είναι οι πόλοι ανάπτυξης και θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και ως προς την χρηματοδότηση. Και μία δεύτερη ερώτηση. Πώς βλέπετε τις τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα μεγάλα προγράμματα. Έχω την εντύπωση ότι τίθεται εδώ ένα θέμα ελέγχου. Επίσης, ε, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τις γνώσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, τι θα κάνουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριο Σάσα Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκαρμεντία για την σημερινή παρουσία της εδώ και να πω το εξής τι αρέσει στον ερευνητή και τι δεν αρέσει. Στον ερευνητή, στην Ισπανία και στην Ευρώπη αρέσει να έχει ασφαλεία στην εργασία του. Δεύτερον, να τον αφήσουν να εργάζεται ήρεμο. Ε, αυτό που δεν του αρέσει είναι η γραφειοκρατία που βιώνει και δεύτερον, ε, ουσιαστικά όλες αυτές οι τεχνοκρατικά εμπόδια που πρέπει να υφίσταται. Αν τα λύσετε αυτά τα προβλήματα θα σας ευχαριστήσουν οι Ευρωπαίοι ερευνητέ ε, να ξέρετε ότι εμείς ε, σας υποστηρίζουμε. Εγώ σας υποστηρίζω. Ευχαριστώ, η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ. Ε, μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ τα μάλλα με το πρόγραμμά σας στον τομέα αυτό. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις ε, που ήθελα να θέσω τέθηκαν. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρώπη προσπαθεί να απαγιωθεί ως μια ε, πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Η Ισπανική Προεδρία σίγουρα θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στον τομέα αυτό, καθώς η στρατηγική της Λισαβόνας φτάνει στο τέλος της τώρα το 2010. Μιλάμε πολύ για μέσα, για διαδικασίες, ε, μιλάμε όμως λιγότερο για τους ερευνητές. Και εδώ ξέρουμε πόσο ε, έχουν αυξηθεί τα επίπεδα επισφάλειας των ερευνητών τα τελευταία χρόνια και παρά τις όλες προσπάθειες η κινητικότητα δεν ήταν επαρκής. Πολλές φορές ε, η κινητικότητα ενισχύει αυτή την επισφαλή τους θέση η Ισπανική κυβέρνηση αποτελεί μία, ένα από τα σπάνια παραδείγματα ε, ανάληψης ε, μέτρων ε, υπέρ των ερευνητών. Ε, μήπως ε, θα μπορούσατε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές που έχετε υλοποιήσει στην Ισπανία να τις διαδώσετε και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο δίκαιο επιστημονικό χώρο που να σέβεται και τα δικαιώματα των ερευνητών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να περιοριστείτε στα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. Καταρχήν, να απαντήσω στην κυρία Γκουτιέρες, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή της. Έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσουμε σημαντικές πτυχές που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση και την λεπίδραση της κατάρτισης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό με τον ίδιο τρόπο που θα προσεγγίσουμε και το θέμα της κινητικότητας των ερευνητών ε, και τις ε, κοινωνικές πολιτικές ε, στο Συμβούλιο Απασχόλησης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε στα πλαίσια των άτυπων συμβουλίων να βελτιστοποιήσουμε την θέση αυτών των πτυχών στο τρίγωνο της γνώσης, στις υπουργικέ διασκέψεις για την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία. Και θα πρέπει να προωθήσουμε αυτούς τους τομείς ε, και νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε προτάσεις σε υπουργικέ συνδιασκέψεις ε, στο περιθώριο, των, στο πλαίσιο με συγχωρείτε, των άτυπων συμβουλίων θα μπορούσαμε να σκεφτούμε επί της αναγκαιότητας ε, αυτών των μέτρων. Τώρα, για, για τις διαφορές που έχουμε μεταξύ διαφόρων μελών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις του ΑΕΠ μας στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ο καλύτερος ε, τρόπος να πείσουμε για περισσότερε επενδύσει είναι να δείξουμε τα αποτελέσματά τους. Εμείς στην Ισπανία ε, ξεκινήσαμε αυτή τη δράση και πραγματικά είναι πολύ αποτελεσματική στην Ισπανία δείξαμε στις μικρές και μεσαίες μας επιχειρήσεις ότι αν επενδύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη αυξάνουν την παραγωγικά τους 16% και 18% την αξία των εξαγωγών τους. Μιλάμε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σε στιγμές κρίσης δημιουργούν θέσεις εργασία πρόκειται για πιο σταθερέ και υφόρες θέσεις εργασία και μάλιστα ε, επιβιώνουν καλύτερα σε στιγμές οικονομικής κρίσης. Εγώ νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και οι επένδυσεις ε, ε, πρέπει να δείξουμε στου πολίτε μα ότι οι επενδύσεις αυτές είναι αποτελεσματικές και ότι οι μεγάλες ε, προκλήσεις αντιμετωπίζονται με την δημιουργία καινούργια γνώσης. Γι' αυτό η κριτική μάζα είναι πολύ σημαντική, η ένωση των κρατών μελών, ε, η ευθυγράμμιση των πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ε, η γνώση για τη γνώση είναι κλειδί, αλλά μιλάμε για άριστη γνώση. Χωρί να έχουμε τομεακού κατακαιρματισμού. Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτά τα δύο θέματα να δείξουμε στους πολίτες μας και αυτό θα πείσει τις χώρες και τους υπουργού οικονομικών μας ότι πρέπει ένα σημαντικό τμήμα του προπολογισμού να εκταμιευτεί για ε, δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Η Ισπανία υπερασπίζει ε, τις ε, περιοχές γνώσης ε, και τη δυναμική που έχουν οι διάφορες περιφέρειες. Είναι ένα τμήμα της διακυβέρνησης αυτό που θέλουμε να το προωθήσουμε που κινούμε τις περιφέρειες. Υπάρχει και ένα τμήμα εμπλοκή τη ευρωπαϊκή επιστήμη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την βελτιστοποίηση των πόρων, αλλά και με τη δέσμευση των κρατών μελών να ευθυγραμμίσουν τι εθνικέ ε, πολιτικέ ε, και τι περιφερειακέ πολιτικέ με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Πρέπει να βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Πρέπει να έχουμε ε, προγράμματα καθρέφτε, αν θέλετε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε πιο αποτελεσματικά πιο γρήγορα με συγχωρείτε στα αποτελέσματα. Και μάλιστα στην Ισπανία είδαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συνοχή μεταξύ των περιφερειών. Τώρα για τη σταδιοδρομία των ερευνητών. Η Ισπανία έχει δεσμευτεί να ε, προωθήσει ε, την ε, στα διαδρομία των ερευνητών και να σεβαστεί τα δικαιώματα των ερευνητών, γιατί όπως είπε και η κυρία Κουτιέρης μόνο έτσι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Οι νέοι που τώρα σκέφτονται τι θα κάνουν στο μέλλον, θα πρέπει να θέλουν να γίνουν ερευνητέ, γιατί το χρειάζεται η Ευρώπη και πρέπει να του ε, προσφέρουμε ένα, ένα ελκυστικό μέλλον, μια σταδιοδρομία που να αναγνωρίζεται κοινωνικά και να ε, βοηθά στην παγίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στην Ισπανία προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά η επιθυμία μας είναι να ε, μοιραστούμε με την Ευρώπη τον αντίκτυπο που είχε στην Ισπανία, το να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα των ερευνητών, ε, τα δικαιώματα κοινωνικής ε, ασφάλισης, να τους δίνουμε υποτροφίες και από την προδιδακτορική ήδη από το προδιδακτορικό στάδιο να δίνουμε υποτροφίες και τελικά να προωθήσουμε και ε, κάποιους τρόπους πρόσληψης ε, των ε, υποψήφιων διδακτόρων. Αυτή είναι η επιθυμία μας και θέλουμε να μοιραστούμε με όλα τα κράτη-μέλη αυτές τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ισπανία σχέση με τα δικαιώματα των ερευνητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις ε, παρεμβάσεις σας και σας ευχαριστώ που μας βοηθήσατε να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή εγκαίρως. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η τελευταία συζήτηση που θα έχουμε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα συνομιλήσουμε αρκετέ φορέ. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα το πρωί και που ήρθατε να μιλήσετε μαζί μα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ε, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα στην αρχή, αλλά η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη δουλειά σας τους επόμενους μήνες.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 Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Σημείο 21, διάλογος πανεπιστημίων επιχειρήσεων, μια νέα εταιρική σχέση. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει μέχρι το μεσημέρι, θα πρέπει να ε, δαπανίσουμε το πολύ 20 λεπτά για κάθε σημείο. Ε, και νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα έχουν πρόβλημα αν ε, ε, αναβάλουμε κάτι για το απόγευμα. Σας παρακαλώ λοιπόν βοηθήστε με. Η κυρία Ριέρα Μαντουρέλη, η πρώτη που θα παρουσιάσει την εκθεσή της, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω για την έκθεση που μόλις ανακοίνωσε ο Πρόεδρος. Και να σας πω ότι αυτό που ήθελα καταρχήν να τονίσω στην γνωμοδότηση είναι ότι το φόρουμ για το διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων είναι καλό μέσο για την εντατικοποίηση της σχέσης ε, μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Και η ενδυνάμωση της σχέσης αυτής είναι ε, σημαντική για να ενισχύσουμε το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή παιδεία, καινοτομία και έρευνα. Αυτό φυσικά θα επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τα ανεπινιστήμια, για τις επιχειρήσεις, για την ανταγωνιστικότητα και τη γνώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαμε επίσης να τονίσουμε ε, στο κείμενο ότι αυτή η σχέση θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Η γνώση και η ενημέρωση μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων θα πρέπει να αφορά και την ε, προσφορά και τη ζήτηση άλλα λόγια, θα πρέπει να μας ε, οδηγήσει όχι μόνο στο να υπάρχει επιχειρηματική κουλτούρα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά θα πρέπει και ε, η πανεπιστημιακή κουλτούρα της γνώσης να εισαχθεί στις επιχειρήσεις, δηλαδή να προωθήσουμε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, πιο επιστημ... αποκαλέσουμε μια επιστημονική επιχείρηση δίνουμε κάποιες ε, ιδέες ε, που θα μπορούσαν να προσταθούν ε, στις προτάσεις της Κομισιόν. Λόγου χάρη, από τη σκοπιά της ζήτησης πιστεύουμε ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε καταρχήν να κάνουν μια καλή διάγνωση των ισχυρών του σημείων σε ό,τι αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση και πώς σχετίζονται αυτά τα ισχυρά σημεία με τις αναγκαιότητες των επιχειρήσεων χωρίς ε, φυσικά να ε, ξεχνούν ε, το θεμελιώδες εκπαιδευτικό τους έργο. Το πρώτο βήμα για την επιτυχία είναι αυτό. Επίσης, τη διαβίβαση της τεχνολογίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις, ε, τα πανεπιστήμια επιφέρουν στην αγορά εργασίας προσωπικό που έχει καταρτιστεί ορθά και είναι καλά προετοιμασμένο, ικανό να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σκοπιά της γνώσης και της αριστείας. Από τη σκοπιά της ζήτησης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησης ε, η μεταμόρφωση ε, της επιστημονικής γνώσης συμμετέχοντας ε, στα ερευνητικά προγράμματα και στα διδακτορικά προγράμματα την ε, πρόσληψη ερευνητών και στη χορήγηση υποτροφιών. Και τα κρατημέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια, να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο που να επιτρέψει μια αυθεντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και να δώσουν και κίνητρα στις ε, επιχειρήσεις έροντας τα διοικητικά εμπόδια δημιουργώντας και μηχανισμούς ε, που να δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στα πανεπιστήμια. Στο έγγραφο της Κομισιόν ε, γίνεται αναφορά επίσης στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ε, νέων διαθρωμένων σχέσεων μεταξύ πανεπιστημίων ε, και επιχειρήσεων. Και σας είπα στην πρώτη μου παρέμβαση ότι αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο σημείο καθώς υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που έχουν γίνει από εμπειρογνώμονες από τις οποίες συνάγεται ότι πιο αποτελεσματική μορφή αυτή τη στιγμή μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων γίνεται μέσω προσωπικών επαφών, ε, μέσω της συμμετοχής σε σεμινάρια και διασκέψεις και μέσω της ε, παροχής ε, υπηρεσιών και έρευνας με σύμβαση. Δηλαδή σημαίνει ότι οι μη διαρθρωμένες μορφές μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές από ότι οι διαρθρωμένες, ή υπερβολικά διαρθρωμένες μορφές συνεργασίας που τελικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα άκαμπτες και μπορεί να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια απλώς σε παροχής ε, υπηρεσιών καινοτομία εις βάρος των ε, ε, επενδυτών ε, ερευνητικών και και εκπαιδευτικών τους ε, δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι μια καλή πρόταση. Βέβαια, αρκεί να γίνεται πάντοτε σε βαστή αυτονομία των πανεπιστημίων και ο χαρακτήρας του δημόσιου ε, ιδρύματος. Επίσης, το STI, οι KICS μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη ε, σχέση. Και για να κλείσω, να πω ότι στην τελευταία παράγραφο θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο αυτού των διαλόγων να ε, υπάρξει αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και όχι μόνο να εντοπίσουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά να ε, εντοπίσουμε και τα καλύτερα φυστάμενα μέσα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό και σε κοινωτικό επίπεδο και Τέλος, ε, βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια αντιδρούν θετικά στα υφιστάμενα κίνητρα που υπάρχουν στα περιφερειακά, εθνικά και κοινατικά προγράμματα για την ε, ανάπτυξη πολιτικών συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία που θα ήθελα να τονίσω στην δική μου έκθεση και Φυσικά, όπως πάντα, είμαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση και σχόλια μπορούν ε, να συνεισφέρουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το σχέδιο γνωμοδότης της κυρίας Μαντουρέλ κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω εξέταση και προώθηση του ζητήματος. Ήδη η κυρία Μαντουρέλ με τη σημερινή της παρουσίαση μας παρουσίασε τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα του θέματος που φέρει, που φέρει για πρώτη φορά ε, σε επαφή δύο διαφορετικούς κόσμους, τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Αυτά όμως πρέπει να συνδεκαστούν, αυτό είναι βέβαιο, το ξέρουμε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων είναι ένα από τα κύρια ζητούμενα καθώς επίσης και η ανάπτυξη μιας ε, ε, επιχειρηματικότερης αντίληψης των πανεπιστημίων ως ιδρυμάτων και όχι ως ατόμων σε σχέση με την αποστολή τους. Τα μοντέλα που σήμερα εφαρμόζονται σε σχέση με τη ε, συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρηματιών περνούν στα περισσότερα κράτη του κόσμου μέσα από τον αντιπρίτανη ε, ε, της Ερευνητικής Επιτροπής και δεν έχει να κάνει με την διαπλοκή του προσωπικού με τις επιχειρήσεις. Η συνεισφορά των επιχειρήσεων τόσο στην αλλαγή του κλίματος αλλά και του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα είναι πολύ σημαντική όπως επίσης η εμπειρία των επιστημόνων στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων, στην επίλυση συγκεκριμένων μέτρων, είναι επίσης εξίσου σημαντική. Οι προτάσεις που ε, κάμω προς την κυρία Μαντουρέλ με την οποία η συνεργασία μου ήταν άριστη θα σας κοινοποιηθούν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου που είναι το deadline. Απλώς η δική μου υπόδειξη είναι ότι θα έπρεπε τα, τα, διδακτορικά προγράμματα να αποκτήσουν μια στενότερη σχέση με τις επιχειρήσεις, ακόμα και με την συμμετοχή προσωπικού από τις επιχειρήσεις στις ε, επιτροπές που επιβλέπουν την εκπόνησή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Καβάλιο. Κυρία Καρβάλιο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με τη γραμματότηση τη κυρία Μαντουρέλ. Θα ήθελα απλώς να κάνω ένα σχόλιο. Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος ε, της αλυσίδα ε, της καινοτομίας, όπω και επιστημονική έρευνα θα έπρεπε να αναπτύξουμε τελικά ε, ένα τομέα εκπαίδευσης για την καινοτομία και η εμπειρία του ΕΕΤ θα μπορούσε να είναι καταλήτης για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις ε, να συμμετέχουν ισότιμα στο καθορισμό των προγραμμάτων στις διαδικασίες δεσκαλίας ε, και ε, στα στάζ. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα πανεπιστημιά μας. Πολλά ε, από τα πανεπιστημιά μας χρήζουν πιο αποτελεσματικά μοντέλα διαχείρισης, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις σταδιοδρομίες, περισσότερη κινητικότητα των ερευνητών και των καθηγητών. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προωθήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων που να δίνει κίνητρα στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ως μέλος ε, της Επιτροπής Προπολογισμών θα ε, προωθήσω Τη δημιουργία ενό προγράμματο προς αυτή την κατεύθυνση για τον εξοχρονισμό των πανεπιστημίων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και καλύτερος διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όλα τα σημεία που άκουσα ε, που αφορούν την έκθεση αυτή αξίζει να τα στηρίξουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να μιλήσουμε για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων χωρίς να ξεχνάμε ότι το βασικό θέμα εδώ είναι η εκπαίδευση. Εκπαιδεύουμε εμπειρογνώμονες του μέλλοντος και ερευνητές του μέλλοντος. Φυσικά, αν λειτουργούν καλά τα πανεπιστήμια, θα εκπαιδεύονται εκεί οι επιρρογνώμονες του μέλλοντος. Ε, και γι' αυτό καλούνται τα πανεπιστήμια να ε, παρέχουν ε, διάφορες δυνατότητες σταδιοδρομίας ε, στους φοιτητές τους. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τα πανεπιστήμια. Ξέρουμε ότι πρόκειται για δημόσια ιδρύματα και δεν γλίτωσαν και αυτά από την οικονομική κρίση στην Ουγγαρία. Απολύθηκαν διάφοροι καθηγητές για να γίνουν περικοπές στις δαπάνες. Τα πανεπιστήμια αυτά λοιπόν δεν μπορούν να προωθήσουν την κινητικότητα με τον τρόπο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καλούνται να κάνουν κάτι, αλλά και οι κυβερνήσεις ε, των κρατών μελών να διαθέσουν ε, πόρους και όπως ήδη υπόθηκε, να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί η κινητικότητα. Τα πανεπιστήμια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τα βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. από την πείρα μου ξέρω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία δημιουργούν την ε, συνοχή, προωθούν τη σχέση ανάμεσα στις ε, επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Καταρχήν ε, θέλουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση ώστε να εκπαιδεύσουμε μηχανολόγους, επιστήμονες κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα πανεπιστήμια. Οι, οι φοιτητές θα μπορέσουν έτσι να ε, διαμορφώσουν την εργασία τους ώστε να είναι θετική και για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να προωθήσουμε τους ερευνητές, αλλά στην ουσία δεν κοιτάμε τι εφαρμόζεται τελικά από τις επινοήσεις ε, των ε, ε, πανεπιστήμιακών. Θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα προώθησης, υποστήριξης, ώστε να διευκολύνουμε την προώθηση της καινοτομίας. Αυτό θα διευκολύνει και τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις να προσεκίσουν ε, αλλήλους. ο κύριος Ροκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνει ο συγκητής να βρει μια εξισορρόπηση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Έχω όμως και δύο δικές μου προτάσεις, δύο προσθήκες. Να πούμε πιο συγκεκριμένα αυτά που είχαμε συζητήσει πριν από τέσσερα χρόνια, εκείνη την ιδέα δηλαδή ότι η γνώση, ας πούμε, να μπορεί να ωφελήσει και κάποια ε, καινούργια επιχείρηση και έτσι να γίνει η σύνδεση με τα πανεπιστήμια. Η πρώτη φάση όλης αυτής της διαδικασίας είναι η σημαντικότερη. Και στις ε, χώρες, στις πρόσφατα ενταγμένες χώρες όπου υπάρχουν οι περισσότερες από αυτές τις καινούργιες επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διάδοση των γνώσεων και η σύνδεση με την έρευνα. Πρέπει όμως να γίνει και δεύτερο στοιχείο που θέλω να προσθέσω είναι ότι για την Επιτροπή μας, η Επιτροπή μας θα έπρεπε να δηλώσει πρώτον ότι υπάρχουν οι γνώσεις, αλλά κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα έχει ταξινομηθεί διεθνώς και πρέπει όλα αυτά να τα γνωρίσουν και οι επιχειρήσεις ε, στη, όπου βρίσκονται, να γνωρίζουν δηλαδή ποια πανεπιστήμια είναι τα καταλληλότερα για αυτές. Εκεί λοιπόν να τα πούμε πιο συγκεκριμένα και να ζητήσουμε από την Κομισιόν τα εργαλεία που διαθέτουμε να τύχουν περισσότερου συντονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπάουερ από την Κομισιόν. Παρακαλώ σύντομα αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν, έχω πολλά να πω. Η, έκθεση αυτή είναι ε, πολύ θετική απέναντι στην πρότασή μας. Ε, συγγνώμη, νόμιζα ότι αυτό είναι το μικρόφωνο. Συγγνώμη. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εσείς επικεντρώνεστε εδώ πέρα κυρίως στην έρευνα. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε και τον ρόλο της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, διότι πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει ε, τεράστιο δυναμικό. Και ε, ε, δυναμικό που μπορεί να επηρεάσει θετικά τις εκπαιδευτικές μεθόδους. Βλέπουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που εφαρμόζουν πολυτομεακή προσέγγιση. Ε, μπορούν να ε, παρέχουν στους ε, σπουδαστές τους πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριέρα Μαντουρέλη έχει να προσθέσει κάτι. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους αλλά και την Κομισιόν για τις παρεμβάσεις τους. Μπορώ να πω μόνο ότι συμφωνώ με όλες τις προτάσεις τους. Τις σημείωσα και περιμένω την αποστολή των τροπολογιών τους. Πιστεύω ότι θα καταρτήσουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Συμφωνώ και με τον καθένα ξεχωριστά θα συζητήσω. Ευχαριστώ. 2 Φεβρουαρίου, η ώρα, περιοθεσμία για τι τροπολογίε ε, και φτάνουμε στην καινοτομία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο συνάδελφος Βίγκλερ έχει το λόγο, ο συζητητής 20 ε, λεπτά παρακαλώ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος ε, ανέφερε ότι πρόκειται για πρώτη ανταλλαγή απόψεων για έκθεση πρωτοβουλίας ε, με θέμα τη γενοτομία σε έναν ε, μεταβαλλόμενο κόσμο. Από το Σεπτέμβριο του 2009 η Κομισιόν ε, στην ανακοίνωσή της ε, ε, αναφέρει τις πρόοδους που έχουν σημειωθεί από το 2005 και αναφέρει και τις δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν στο μέλλον. Η καινοτομία προέρχεται από τις επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές. Επικροτούμε την ανακοίνωση και εδώ ισχύει ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της εάν οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ε, γενικά πάντως η ανακοίνωση αυτή παραμένει στην επιφάνεια των ε, πραγμάτων. Η κρίση ε, των προόδων που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι θετική και αναφέρεται στην πράξη καινοτομία στο Innovation Act, το οποίο προβλέπεται το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για τον Μάρτιο-Απρίλιο φέτος. Είναι ε, πηγόντως απαραίτητη μια καλύτερη στρατηγική. Ε, η στρατηγική καινοτομία ε, θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η απασχολησιμότητα, το, ε, η αλλαγή του κλίματος ε, κλπ. Ε, στόχοι που συνδέονται με την στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Η Κομισιόν λοιπόν αναφέρεται ε, στην μελλοντική πολιτική καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, θα θέλαμε να την σχολιάσουμε. Η πρώτη μου ερώτηση προς τους εκπροσώπους της Κομισιόν. το πότε μπορούμε να υπολογίζουμε να λάβουμε το σχέδιο δράσης για την πολιτική καινοτομία, πώς θα ληφθούν υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου και ποια θα είναι η σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία του ε, εγγράφου που θα εκπονήσω. Η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να είναι ευρεία και θα πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους ε, ε, τομείς της καινοτομίας και σε αυτούς που δεν συνδέονται με την τεχνολογία. Για παράδειγμα στις υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζεται το δυναμικό και όσον αφορά τις διαδικασίες και όσον αφορά τα προϊόντα και θα είναι ένα θέμα το οποίο θα επηρεάσει πολύ την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, χημεία, ε, παροχή ενέργειας, αυτοκίνητα, αεροπλοεία, το διάστημα κλπ. Η καινοτομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο για ε, εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στους ε, τομείς που ηγείται να ε, αναπτύξει ακόμα περισσότερο τον ηγετικό της ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε τα ισχυρά μας σημεία. Πολύ συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει τα κλάστερ γνώσης των κρατών μελών ε, ε, ώστε να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο και στο μέλλον. Και θα πρέπει ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ε, τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις καινοτομίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται αέρα να εισπνέουν για να μπορούν να είναι καινοτόμε. Ε, θα πρέπει να έχουν καλές συνθήκες. Θα πρέπει να ε, ελαφρύνουμε το ε, γραφειοκρατικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό έχει να κάνει με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, στατιστικών στοιχείων κλπ. Επίσης θα πρέπει να παράσχουμε καλύτερες συνθήκες ε, όσον αφορά τα ε, επενδυτικά κεφάλαια κινδύνου θα πρέπει να ε, τα δούμε όλα αυτά υπό το φως της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που θα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Είμαι διατεθειμένος με την ανταλλαγή απόψεων σήμερα να ξεκινήσω να λαμβάνω ε, διμερώς προτάσεις από την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για να εκπονήσουμε την έκθεση αυτή η οποία είναι τόσο σημαντική για το μέλλον ε, όσον αφορά τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα ε, θα τα αναφέρει ο Πρόεδρος. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σιμάνσκι razy e, e, wracamy do tematu polityki innowacyjnej, tyle razy natrafiamy na jeden podstawowy problem. E, επαναρχόμαστε συνεχώς στο θέμα της έρευνας και ανάπτυξης και πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, την κακή χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη ε, σε σύγκριση με τις ε, χώρες που ηγούνται στον τομέα, ε, με τις άλλες χώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία λύση, διότι τα διάφορα κράτη έχουν ε, διαφορετικές ε, θέσεις. Και ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις επιχειρήσεις. Μπορούμε όμως να προστατεύσουμε καλύτερα τη διανοητική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Εάν δεν εξαλείψουμε το πρόβλημα αυτό, αυτό θα στοιχήσει πολύ στην Ευρώπη και στο μέλλον δεν θα υπάρχει η ευκαιρία να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις. Ε, το ε, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρυστεχνίας μάλλον είναι κάτι υπερβολικά φιλόδοξο. Δεν έχουμε βρει λύση ακόμα. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να ε, επικεντρωθούμε περισσότερο στην αμοιβαία αναγνώριση των διπλωματών ευρυστεχνία και να ανοίξουμε μια συζήτηση όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης καθώς ε, και ε, να σκεφτούμε τη χρηματοδότηση της μετάφρασης, ε, της μεταφοράς των διπλωμάτων έβρεση τεχνίας. Νομίζω ότι το, η λύση εδώ είναι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η κυρία Χέρσογκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω καταρχήν αντικαθιστώντας την κυρία Μέρκες που δεν μπορεί να παραστεί και έπειτα και εξ μου. Δύο ερωτήσεις έχω προς την Κομισιόν. Θα μπορούσε να μας δώσει μια αξιόπιστη απάντηση για το χρονοδιάγραμμα του νομοσχεδίου καινοτομία Innovation Act και θα μπορούσε να μας δώσει μερικές περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το πρόγραμμα δράσης που το συνοδεύει για τη σκιώδη δε εισηγήτρια θέλω να έχω την απάντηση να τη τη μεταφέρω. Τώρα, εξ ονόματός μου, ως πρώην εισηγήτρια για το νομοσχέδιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επειδή με ενδιαφέρει και αυτό το θέμα και η καινοτομία και το συζητώ εδώ στο Κοινοβούλιο, ασχολούμαι με αυτό στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό, θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο το νομοσχέδιο των μικρομεσαίων ήταν πολύ καλή πρωτοβουλία, αν και έχω απογοητευτεί με αυτά που διάβασα εδώ στην στο πρόσφατο έγγραφο για την καινοτομία. Μπορούν να υπάρξουν και πολλές βελτιώσεις. Για μένα η καινοτομία ορίζεται ως περισσότερη αποτελεσματικότητα με καλύτερη χρήση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η καινοτομία δεν είναι κυρίως τεχνικό θέμα, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις ευκαιρίες που έχουμε ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών για καινοτομία και στα καινούργια επιχειρησιακά πρότυπα. Υπάρχει χώρος για βελτιώσεις για την επόμενη δεκαετία. Παραδείγματο χάρη βάση των ψηφιακών εξελίξεων που μας δίνουν τελείως νέα βάση για να προχωρήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης του εγγράφου και αυτός είναι και ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, Άλλα δύο ερωτήματα. Ενισχυμένη συνεργασία θα θέλαμε να υπάρξει μεταξύ γενικών διευθύνσεων, επιχειρήσεων και έρευνας, διότι η καινοτομία δεν είναι απλώς έρευνα, είναι και η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς σχεδιάζετε λοιπόν να συνδυάσετε τη δουλειά των δύο γενικών διευθύνσεων για να μην υπάρξει κατακαιρματισμός. Η κυρία Καβαρβάλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η καινοτομία στην Ένωση πρέπει να μπορέσει να λύσει τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα διατυπώσω ορισμένες συστάσεις. Πρώτον, η αλλαγή του κέντρου βάρους από, την τεχνολογ... από τις τεχνολογικές αλλαγές στις κοινωνικές αλλαγές. Πρέπει να φύγουμε από το αυστηρά τεχνικό πρότυπο σε, μια, σε ένα πιο ευρύτερο ορισμό που να συμπεριλαμβάνει και τις κοινωνικές καινοτομίες και τις καινοτομίες της κοινωνικές υπηρεσίες. Δεύτερον, η επιστήμη και η καινοτομία δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν κενό. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες όπως η κινητικότητα, το ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομία, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ ειδικών επιστημόνων, δηλαδή η κατάργηση φραγμών. Και βέβαια ανοιχτός ανταγωνισμός στην καινοτομία. Τρίτον, περισσότερες δαπάνες για την έρευνα αφού έχει δυσκολίες δε ο δημόσιος τομέας γι' αυτό να χρησιμοποιηθεί ο ιδιωτικός μέσω ιδιωτικής συγχρηματοδότησης, φορολογικής πολιτικής, βαρακινδυνευμένων κεφαλαίων κλπ. Και τρίτον, καλύτερος συνδυασμός καινοτόμων προγραμμάτων ή προγραμμάτων καινοτομίας μεταξύ των χωρών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την συμφωνία μου με όσα ακούστηκαν, ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία που πρέπει να λάβει η Επιτροπή μας και διότι αυτό δείχνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε αποτελέσματα στην πολιτική και των χωρών μελών για τα θέματα της καινοτομίας. Η κυρία Κουίν μας είπε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός από την Κομισιόν. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό ώστε να εξελιχθούν τα πράγματα γρήγορα πριν το καλοκαίρι. Και έπειτα από λίγο πιο νομική άποψη να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε στη συζήτηση γιατί το θέμα είναι πολύ ευρύ και αν βασιστούμε στα έγγραφο της Κομισιόν ε, πριν από τέσσερα χρόνια δεν θα μας αρκέσει αυτό γιατί από τότε άλλαξαν τα πράγματα. Η Ισπανική Προεδρία ίσως θα έπρεπε να ζητήσει μια αλλαγή να μην κάνουν πλέον τα κράτη-μέλη ό,τι θέλουν στο θέμα της έρευνας και της καινοτομίας γιατί δεν είναι αυτό αποτελεσματικό και δεν πρόκειται να οδηγήσει στην Ευρώπη του 2020 που θέλουμε. Θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα γενικά. Τώρα, αν αυτό απαιτεί έκθεση πρωτοβουλίας ευρεία, βάσης ή επικέντρωση στα βασικότερα, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Και το τονίζω, αυτό αφορά ιδιαίτερα την Κομισιόν. Από την Κομισιόν ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι. Να σα κάνω ορισμένε αποσαφηνήσει καταρχήν για τα διαδικαστικά. Έγινε λοιπόν η ανακοίνωση αυτή της Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά οργανώσαμε μεγάλες διαβουλεύσεις για να έχουμε πληροφορίες ως προς το, τις απόψεις των ενδιαφερομένων που τώρα τους λέμε stake και holders. Έτσι ώστε να έχουμε μία όσο δυνατόν ευρύτερη πληροφόρηση για το τι συζητιέται στην Ευρώπη από τους ενδιαφερόμενους ή stakeholders. Ο κύριος Μπαρόσο βέβαια καθόρισε ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης και υπάρχει μια στρατηγική για το 2020 που θα δημοσιευθεί σε λίγες εβδομάδες. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο λοιπόν των guidelines του κυρίου Μπαρόζου θα καθορίσουμε αυτή τη στρατηγική EU 2020. Και τώρα για να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορέσει να εγκριθεί τον Απρίλιο όπως είχαμε προβλέψει αρχικά. Μάλλον Ιούνιο με Σεπτέμβριο το βλέπω. Δεν μπορώ να το προδικάσω βέβαια γιατί εξαρτάται από τη δραστηριότητα της μελλοντική Επιτροπής. Αν νομίζω πιο λογικό είναι να φανταστούμε για να μπορέσουν και ο κύριος Σταγιάννη και η κυρία Γκριν να προετοιμαστούν καταλήλως να προβλέψουμε έγκριση μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Για τη συνεργασία μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων Έρευνας και Επιχειρήσεων, εγώ είμαι από τις επιχειρήσεις και η Γενική Μονάδα για την Καινοτομία ε, συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση της Έρευνας. Έχουμε επαφές, οι οποίες μάλιστα θα γίνουν εντατικότερες τις επόμενες εβδομάδες, γιατί αυτό το πρόγραμμα καινοτομία είναι σημαντικό στρατηγικό σχέδιο και για την έρευνα και για την καινοτομία. Εμάς η προσέγγιση μας είναι σαφής. Θεωρούμε ότι είναι η έρευνα πολύ σημαντική για την καινοτομία, αλλά ότι την τελευταία αυτή πρέπει να τη θέσουμε νέας βάσεως, δηλαδή πιο ευρύτερα να τη δούμε, διότι η εμπειρία μας δείχνει ότι η τεχνική και το design όπως και η εφαρμογή νέων επιχειρησιακών προτύπων ή business models δείχνουν ότι η καινοτομία έχει εξελιχθεί με το χρόνο ως έννοια. άκουσα με προσοχή όλα τα σχόλια των Ευρωβουλευτών και γενικά συμφωνούμε με την προσεγγίσεις τους. Και θα λάβουμε τα κατάλληλα μαθήματα από αυτά που μας είπατε. Καταρχήν δεν πρέπει να γνωρίσουμε τη σημασία που έχει η τεχνολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο και τη σημασία που δίνουμε σε αυτήν. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα νέα εργαλεία όπως τα κλάστερ και τα lean market για την καινοτομία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο φαντάζομαι ότι μπορώ να σταματήσω εδώ και αν θέλετε αποσαφηνήσεις να μου τις ζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ. Θέλετε πάλι το λόγο, όχι. όχι. Τότε το από αποτέλεσμα είναι ότι δεν βρισκόμαστε υπετρομερή χρονική πίεση, αλλά όσο πιο νωρί ε, παρουσιάσουμε την έκθεσή μα, τόσο ε, καλύτερε δυνατότητε έχουμε να επηρεάσουμε τι εργασίε ε, στην Κομισιόν. Δηλαδή, καλό θα είναι να λάβουμε απόφαση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Ζήτω συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενο θέμα, επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή εντό τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η κυρία Βαλεάν. Well, uh, thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι, υποδο... οι ενεργειακές υποδομές και η συλλογή στοιχείων για αυτές για την ε, κατάστρωση μια στρατηγικής είναι το θέμα μας. Υπάρχει πρόταση AIMS για τις πιθανές εξελίξεις στις ενεργειακές υποδομές ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ανάλυση των προοπτικών για τη διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς γενικότερα και για την εφαρμογή μιας πανενωσιακής ενεργειακής πολιτικής. Έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των συντακτών τους. Όλοι θέλουμε να καταλήξει η Κομισιόν σε μια σωστή ανάλυση Υπάρχει βέβαια ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των στοιχείων που χορηγούν οι επιχειρήσεις, της προέλευσης τους δηλαδή. Για να επισέλθω όμως στην ουσία, θα αρχίσω από το θέμα του νομικού υποβάθρου. Οι συνάδελφοι ζήτησαν αλλαγή από το 100, στο 194 τη συνθήκη τη Λισαβόνα, εννοώ για την ενεργειακή πολιτική. Η νομική επιτροπή θα ψηφίσει τώρα για το θέμα αυτό και από ό,τι ξέρουμε θα υποστηρίξουν την αλλαγή αυτή του νομικού υποβάθρου η οποία θα δώσει στο Κοινοβούλιο δικαιοδοσίες απόφαση. Το Συμβούλιο δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένο όμως να συμφωνήσει και γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σας για να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή ακόμη και αν χρειαστεί να πάμε στο δικαστήριο. με βάση τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί συζήτησα και εγώ με τους σκιώδεις για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Γενικά υπάρχει υποστήριξη των συναδέλφων από το συμβιβασμό 5 για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών. Η Κομισιόν υποχρεώνεται να, υποχρεω... να δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές όπως λέει ο συμβιβασμός 6, η συμβιβαστική 6. Και στο συμβιβασμό 7 αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Αυτό που ακόμη εκκρεμεί και πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω είναι το, η χρονική στιγμή κατά την οποία θα υποχρεώνεται, θα γίνεται υποχρεωτικά η πληροφόρηση, η χορήγηση των πληροφοριών. Αν δεν είναι υποχρεωτική η στιγμή αυτή, τότε ο, υποχρεω... ο εμπιστευτικός χαρακτήρας γίνεται κάτι το αρνητικό. Οι πληροφορίες που δίνονται στην Κομισιόν πρέπει να είναι πληροφορίες που έχουν ήδη χορηγηθεί στα κράτη-μέλη. Αλλά ο εμπιστευτικός χαρακτήρας σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος σεβασμού και των διατάξεων κατά των τραστ και μονοπωλίων. Υπάρχει και ένα πρόβλημα ως προς το τι θα προβλεφθεί νομικά για την πληροφόρηση και των ε, εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων ως προς τον καθορισμό της, επιχειρησιακής, της πολιτικής της επιχείρησης όταν γίνεται η χορήγηση των πληροφοριών. Ίσως ένας τρόπος είναι να είναι πολύ μικρή η διορία από τη στιγμή που θα είναι υποχρεωτική χορήγηση μέχρι την εφαρμογή ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αμβεβαιότητα για τους εργαζόμενους. Και εδώ θα μπορούσε να υπάρξει ένας συμβιβασμός ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη που έχει η Κομισιόν να γνωρίζει τα στοιχεία αυτά με την ακρίβεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες θα προσπαθήσω να κρατηθούν οι χρησιμότερες για την Κομισιόν και θα φροντίσω βέβαια να κρατήσω όσες είναι σωστότερες τεχνικά, όσες συμφωνούν με τους στόχους του κανονισμού και δεν αλλάζουν το κέντρο βάρους ή δεν ξεφεύγουν από το θέμα. Ξέρουμε ότι όλοι έχουμε αυτό τον πειρασμό να καταθέτουμε τροπολογίες εκτός θέματος. Χρειάζεται λοιπόν ακόμη λίγη δουλειά, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί σχεδόν όλων και για την ψηφοφορία που προβλέπεται για την επόμενη πέμπτη. Θα ακούσω τώρα τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαντό. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την καλή δουλειά που έγινε για το συντονισμό. Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητικό το έργο της κυρίας Βελέαν. Κάτι πολύ σημαντικό που διακυβεύεται εδώ έχει να κάνει με την πώς μπορούν να παρουσιαστούν τα ενεργή ενεργειακά μας ε, σχέδια. Και εδώ πρέπει να εξεύρουμε την απαραίτητη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και να τη συμφιλιώσουμε αυτή με το να μην αμφισβητήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέσων. Αν ε, δεν ε, έχουμε πάρα πολύ χρόνο για την κοινοποίηση, τότε από είναι εμφανές δεν θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τις επενδύσεις που έχουν προβλεφθεί. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε διδασμό για το θέμα αυτό. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες ε, και ουσιαστικές λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιώσουμε. Όμως υπάρχει κάτι σημαντικό επί το οποίο θέλω να επιμείνω όλες οι υποδομές που σχετίζονται με αποκεντρωμένους ε, τύπους ε, ενέργειας ε, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που έχουμε προτείνει. Μας μας φαίνεται σημαντικό κάθε, όχι να υπάρχει κοινοποίηση κάθε μικρού έργου, αποκεντρωμένου έργου ενέργειας, αλλά η Κομισιόν να μπορέσει να αποκτήσει τα εθνικά σχέδια για αποκεντρωμένης ενέργειας έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μία πλήρη εικόνα για τις ε, ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης. Χθες Στη συνεδρίαση με την κυρία Βελεάν και με το σκιώδη σογητή συζητήσαμε την αναγκαιότητα να συμπεριλάβουμε τις ενεργειακές υποδομές που μπορεί να βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που ε, τροφοδοτούν ε, καταρχήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενφερθήκαμε στο ένα παράδειγμα, ε, χάρη ε, όταν έχουμε τέτοιες ενεργειακές υποδομές, ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υποδομές που συνεισφέρουν στην προσφορά ενέργειας για την Ευρώπη. Κ. Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, στόχος αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης έχει να κάνει με την καλύτερη εναρμόνιση των ε, σχεδίων. Ίσως ε, ακόμη να μην μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, δυστυχώς, αλλά ε, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για προτεραιότητες με ενεργειακούς όρους. Έχουμε εδώ και το στοιχείο του ανταγωνισμού που μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των εθνικών διαδικασιών και να προωθήσει τις διασυνδέσεις. Συγγνώμη κύριε Γκέρεκ, υπάρχουν προβλήματα μετάφρασης. Από ποια γλώσσα, αγγλικά, είχαμε πρόβλημα στα αγγλικά. Μπορούμε να ελέγξουμε αν λειτουργεί η αγγλική καμπίνα, λειτουργεί καλά η διερμηνία. Στα αγγλικά υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης, λέει ο Πρόεδρος. Είναι καλύτερα τώρα που θα πρέπει να μιλάω, γιατί αλλιώ δεν έχετε και τι να μεταφράσετε. Αγγλικά, ακούγονται τα αγγλικά, όχι ακόμα. Ακούγονται τα αγγλικά. Τα γερμανικά ακούγεται, ακούγονται. Ωραία, πάμε πάλι. Να δοκιμάσουμε πάλι. Από την αρχή λέει ο μιλητής όχι. Λοιπόν, για να διατηρήσουμε τη συνοχή και να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Αυτές οι υποδομές θα πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια και ουσιαστικά αυτό είναι το περιεχόμενο των τροπολογιών μου. Ζητώ συγγνώμη σε όποιον έχει διαβάσει τις τροπολογίες μου, όμως ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας πλήρης ορισμός ακόμη ε, για τις υποδομές Δηλαδή γίνεται λόγος λόγου χάρη για ραδιενεργά απόβλητα, για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και η δική μου τροπολογία 36 μπορούσε να έχει να κάνει με τα απόβλητα, όπως θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλα είδη αποβλήτων, όπως το χάρη βιομάζας, διοξίδου του άνθρακα ή ραδιενεργών αποβλήτων. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα πολύ πλήρη ορισμό εδώ. Ε, και η τροπολογία μου 77 μιλά για όλη τη διαδικασία αποθήκευσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική μια άλλη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Αν δούμε όλες τις τροπολογίες και τις ε, αναλύσουμε, δεν ε, υπάρχει εδώ ένα σύστημα ε, το οποίο ουσιαστικά να καλύπτει όλες τις ενεργειακές υποδομές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρνέσκο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βαλάν, Βαλάν δηλαδή, που δέχτηκε και τις τροπολογίες μας για την εξέβρεση συμβιβασμού. Η ομάδα μου υποστηρίζει τις συμβιβαστικές τροπολογίες και θεωρούμε ότι το τελικό κείμενο θα μπορέσει να εγκριθεί εύκολα. Θα ήθελα να επιμείνω μόνο επί ορισμένων σημείων που απομένουν εκρεμή. Η Κομισιόν πρέπει να συντάξει έκθεση ως προς την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης. Και αυτό πρέπει να το κάνει κάθε δύο χρόνια διαθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τηρεί απόρριτο το χαρακτήρα, την προέλευση δηλαδή των πληροφοριών από τις διάφορες επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να εξετάσουμε με τι μορφή θα κάνει τη δημοσίευση αυτή. Εμείς θα θέλαμε να είναι συνδυασμένα δεδομένα ε, ε, στο εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, για να μπορέσει να κρατηθεί απόρριτος ο χαρακτήρας των εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να ζητηθεί από ορισμένε επιχειρήσεις ενεργειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό ζητούμε να είναι συνδυασμένα τα στοιχεία για να φαίνεται καθαρά η παρουσίασή τους. Στο κείμενο λέει specific body και θελήσαμε να κάνουμε έναν ορισμό της έννοιας αυτής για να δούμε γιατί specific bodies πρόκειται για οργανισμούς δηλαδή που θα χορηγούν αυτά τα στοιχεία ή που θα κάνουν την ανάλυση μάλλον. Θα θέλαμε επίσης να υπάρχει κάποια συνέχεια ή παρακολούθηση των σχεδίων επένδυσης στην ενέργεια των χωρών μελών είτε από κράτη είτε από επιχειρήσεις τρίτες που έχουν όμως επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, τρίτες, εφόσον αυτά έχουν επίπτωση στην ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. Τέλος. Κρατήσαμε την έκφραση low carbon, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας στο ΕΛΚ και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Ευχαριστώ για την Κομισιόν, ο κύριος Ρίπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον της ε, στην πρόταση αυτή και ιδιαίτερα την κυρία Βαλεάν για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην προσπάθειά της να συνδυάσει το μεγάλο αριθμό προτάσεων σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Διότι για 10 άρθρα έχουμε σχεδόν 140 τροπολογίες. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάποιο συνδυασμό τους και είμαστε ευγνώμονες για την, τις προσπάθειες της κυρίας Βαλέαν. Οι περισσότερε τροπολογίε επί τη ουσία ε, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Κομισιόν. Ε, σκέφτομαι ε, το θέμα τη κοινοποίηση, τι θα πρέπει να γίνεται με τι πληροφορίε που συλλέγονται στι αναλύσει όσον αφορά τη διαφάνεια, τα όσα υπόθηκαν για την εμπιστευτικότητα. Και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, επικροτούμε την επέκταση ώστε να καλύψει και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και επίσης σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να δεχτούμε τα κατόφλια που προτείνονται. Σήμερα το πρωί μόλις είδαμε το κείμενο των συμβαστικών τροπολογιών και διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση ότι Η πενταετία πριν ξεκινήσουν οι επενδύσεις διατηρείται, διότι υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για το θέμα αυτό. Πάντως μπορούμε να δεχτούμε τη συμβεστική τροπολογία με τη φορφή που έχει τώρα. Ε, εκεί που ανησυχούμε λίγο περισσότερο είναι η περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογής ε, που ξεπερνάει αυτά τα σημεία που ανέφερε, που θα αυξήσει το γραφειοκρατικό άχθος και ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό λίγο πιο προσεκτικά. Επίσης θέλουμε να αποφύγουμε ο κανονισμός αυτός να ε, γίνει ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται και με άλλη δευτερογενή νομοθεσία. Γενικά λοιπόν είμαστε ευγνώμονες. Μπορούμε να δεχτούμε πολλές από τις ιδέες που προβάλλεται. Θα προσπαθήσουμε να τις εισάγουμε στην συζήτηση στο Συμβούλιο, ώστε να συμπεριληφθούν στο βαθμό που είναι δυνατό και εκεί. Όσον αφορά τη νομική βάση, έχουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας μας και ο, ο Επίτροπος Πίπαρξ έχει ε, αναφέρει ότι ε, τα άρθρα 137 και 187 της συνθήκης είναι ε, το, η απαραίτητη νομική βάση. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τι προτάσει στο κείμενο του Συμβουλίου στον βαθμό που είναι δυνατόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Βαλιάρ και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μία σύντομη παρέμβαση από τον κύριο Μπάλσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτος είχα ζητήσει το λόγο. Μία ερώτηση. Μοιράστηκαν εδώ συμβιβαστικές προτάσεις. Θα ψηφίσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ή όλες τις τροπολογίες που βρίσκονται στο μεγάλο φάκελο. 4 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και έτσι καταπίπτουν οι βασικές τροπολογίες της πρότασης αυτής. Θα υπάρξει κατάλογος τότε, όχι σήμερα όμως. Στις 4 Φεβρουαρίου θα υπάρξει πρόταση όταν ε, εγκριθούν δηλαδή οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα υπάρξει σχετικός ε, κατάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Να πω όμως τότε ότι συμφωνώ με τις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά δεν συμφωνώ, διότι τα πράγματα με τα οποία διαφωνώ δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ε, συμβαστικές τροπολογίες, οπότε όλα είναι εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια, να επιβεβαιώσω ότι έχω λάβει επιστολή από τον Επίτροπο Πίμπαλξ όσον αφορά τη νομική βάση. Η νομική υπηρεσία συμφωνεί με την δική μας θέση όσον αφορά τη νομική βάση. Αυτό είναι ίσως ενδιαφέρουσα σημαντική, ε, ε, ε, ε πληροφορία για τους συναδέλφους. Η κυρία Βαλεάν, θέλετε πάλι το λόγο. Κυρία Βαλεάρ, να κάνω κάποια σύντομα σχόλια για όσα είπαν συνάδελφοι. Δύο φορές ε, προέκυψε ιδέα του να συμπεριληφθούν ε, και εταιρείε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ διαφωνώ ως θεμαρχής. Καταρχήν, γιατί έχουμε το θέμα της εξοδοφικότητας, αλλά και δεύτερον γιατί σχετίζονται με τον κανονισμό μόνο αν ε, υπάρχουν υποδομές που θα πρέπει να εισάγουν την ενέργεια στην Ευρώπη και υπάρχει κοινοποίηση για αυτές οι υποδομές συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο που εγώ θα πήγαινα παραπέρα. Και επίσης ε, υπάρχει ένα θέμα με το, ε, πολλαπλούς ορισμούς με πολλούς ορισμούς, πρέπει να αποφασίσουμε αν, όπως είπε ο κύριος Γκέικ, ε, πρέπει να ορίσουμε την υποδομή και να πάμε τόσο μακριά και να ακολουθήσουμε δηλαδή το πνεύμα τροπολογιών ή να το αφήσουμε για μια άλλη φορά. Από ό,τι καταλαβαίνω από την Κομισιόν, ο στόχο αυτού του νομοθετηματό δεν είναι να τροποποιήσει τις επενδύσεις. Δηλαδή, το θέμα αυτό να ξέρουμε τι γίνεται προκειμένου να τροποποιηθούν οι επενδύσεις δεν είναι κάτι αποδεκτό από μένα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν, όμως το Φεβρουάριο τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα την λευκή βίβλο της Κομισιόν για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Καταρχήν η συντάκτρια Ματίας, η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορώ να πω ότι η πορτογαλική μετάφραση λειτουργεί πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να συγχαρώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω τώρα να λάβω τα σχόλιά σας πέρα από αυτά που έχω λάβει ήδη. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή. Πιστεύω ότι η εκπόνηση μιας λευκής δίβλου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι πάρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στο πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Είναι προφανές ότι κάθε φορά πρέπει να ενισχύουμε περισσότερο τη συνεργασία ότι μιλάμε εδώ για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά έχει και διαφοροποιημένες επιπτώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το έγγραφο επικεντρώνεται κυρίως στα μέσα προσαρμογής, όμως είναι δύσκολο ε, να διαχωρίσουμε το θέμα αυτό από τα μέτρα μετριασμού. Έτσι λοιπόν κάποιες από τις προτάσεις που γίνονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να, αναλάβουμε προσπάθειες για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, αλλά εγώ κάνω πολύ συγκεκριμένε προτάσεις σε σχέση με τους ε, τομείς ε, που φύγονται εδώ, δηλαδή την ε, έρευνα στον τομέα της ενέργειας λόγου χάρη. Αυτές τις προτάσεις κάνω για την Κομισιόν σε αυτού θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία γιατί έχετε διαβάσει το έγγραφο, έχετε προσβεστεί το έγγραφο, απλώς θέλω να τονίσω κάποια σημεία σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τις υποδομές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες συνέπειες στις υποδομές και επομένως στο ε, σχέδιο του ανεφοδιασμού αλλά και στο σχέδιο των υφιστάμενων υποδομών. Το κόστος θα είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τα μέτρα προσαρμογής που θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μια πρώτη έκκληση λοιπόν κάνω στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη να προβλέπουν στα εθνικά του σχέδια δάση ε, τη χορήγηση πληροφοριών όχι μόνο για αυτό το κόστος αλλά και για την κατανομή του κόστους. Ένα δεύτερο σχόλιο, ε, να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα να συμπεριλάβουμε νέα μέτρα σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, ε, προκειμένου να ενισχύσουμε την ασφάλεια αλλά και τη χρήση της παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τα εναρμονισμένα μοντέλα για την ε, κατασκευή και που προβλέπονται ήδη μέσω του Eurocodes. Παραδείγματο χάρη έχουμε την νομοθεσία για τα νέα κτίρια, νομοθεσία για ε, την αξιολόγηση, περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Νομίζω ότι πρέπει να διαρθρώσουμε τους τομείς αυτές. Ένα τρίτο σημείο έχει να κάνει με τον ενεργειακό εφοδιασμό. Νομίζω ότι πρέπει να ε, τονίσουμε ότι αυτές οι διατάστασεις πρέπει να τις ε, θεωρούμε από μια σκοπιά αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και πέρα από την αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει σε μια αλλαγή στην ε, καθολική πολιτική, παγκόσμια πολιτική ενεργειακής αποδοτικότητας, δηλαδή να ενισχύσει την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η οδηγία του 2009 και καλύτερα κρατημέλη μελη να υποβαίνουν μέχρι τις 30 ε, Ιουνίου 2010 τα εθνικά σχέδια δράσης. Το τέταρτο σημείο έχει να κάνει με την αγκαιότητα να ε, ενισχυθούν οι ιδιωτικέ όσο και οι δημόσιες επενδύσεις ε, και σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωσης και σε επίπεδο κράτους μέλους. Εκεί έχω κατά νου την η κρατική συνεργασία και τα εθνικά σχέδια δράσης ε, που έχουν να κάνουν με την έρευνα ε, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείο 5. Να λάβουμε υπόψη ότι οι κλιματικές αλλαγές ε, έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και επομένω υπάρχει αναγκαιότητα να διατεθούν οι πόροι για την προσαρμογή αυτή και οι πόροι αυτοί δεν θα πρέπει να περιοριστούν ε, στα χρήση των εισόδων από το σύστημα εμπορίας ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θέσουμε και στη Λευκή Βίβλο. Έκτον ε, και σχεδόν κλείνω. Να πούμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα τομέα έχουν συχνά συνέπειες και σε άλλους τομείς. Καταρχήν, ενίσχυση των δημόσιων πόρων στο πλαίσιο της διεθνής έρευνας και στο πλαίσιο του 8ου προγράμματος πλαίσιο που προετοιμάζεται τώρα. Αυτό είναι ένας ε, τομέας ε, που πρέπει να έχουμε διεθνή συνεργασία. Ο άλλος τομέας έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των ε, χρηματοοικονομικών πόρων και τη χρησιμοποίησή τους στην έρευνα και στην ανάπτυξη διοχέτευσή τους ε, αυτή πρέπει να γίνει μέσω πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η Κομισιόν ε, και τα κράτη-μέλη μέσω ενός ε, παγκοσμίου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Και κλείνω αναγνωρίζοντας τη σημασία των πρωτοβουλειών σε τοπικό επίπεδο ε, ως τμήμα της, ε, του αγώνα και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Όπως ε, σας είπα λοιπόν, είμαι διαθετημένη για να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και στο μέτρο του δυνατού να τα συμπεριλάβω στην χρηματοδοτησή μου. Ευχαριστώ. Bedanke mich herzlich. Dann haben die σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουν τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι Σκιώδης και άλλοι. Ποιος, ζητάει το λόγο. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θεωρούμε ότι χρειάζεται ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία και ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση τις προσαρμογές είναι κάτι το τελείως απαραίτητο. Επίσης συμφωνώ με την συγκίτρια για την αναγκαιότητα εθνικών σχεδίων προγραμμάτων δράσης. Οι ενεργειακές υποδομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές αλλά και ευάλωτες, ευαίσθητες και γι' αυτό πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες μελέτες κόστους-οφέλους. Τώρα, αλλιώς το κόστος θα αυξηθεί. Ε, και επ' αυτού συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι η γνωμοδότηση μας πρέπει να βασίζεται επίσης και να δίνει μεγαλύτερη προσοχή δηλαδή στα θέματα που είναι δικής μας δικαιοδοσίας όπως οι προσαρμογές όπως λέει και η έκθεση εδώ μάλλον το σχέδιο γνωμοδότησης ε, λείπουν αυτά πρέπει να δείξουμε ότι οι υποδομές είναι ευαίσθητες γενικότερα και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές που είναι σημαντικότερες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον ενεργειακό τομέα βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά υπάρχει και ο τομέας των μεταφορών η σημασία που έχουν οι κλιματολογικές αλλαγές, οι επιπτώσεις τους έχουν, είναι σημαντικές και για τους σιδηροδρόμους ας πούμε. για τη συντήρηση ή την κατάσταση του υλικού. Ε, ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι τηλεπικοινωνίες, επηρεάζονται από τέτοια φαινόμενα. Και κάτι άλλο οι κλιματολογικές αλλαγές επηρεάζουν γενικότερα τη βιομηχανία αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη οι πλημμύρες. Άμα δεν υπάρχει υποδομή αντιμετώπισης πλήττουν και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να δούμε τι πρότυπα εφαρμόζονται και αν χρειαστεί να βελτιωθούν και να προβλεφθούν μέτρα αντιμετώπισης και από τις επιχειρήσεις καθώς και ανάπτυξη ε, δημοσιονομικών υπηρεσιών που να χορηγούν εγγυήσεις στους επιχειρηματίες, στις ασφάλειες δηλαδή. Επίσης να τονίσουμε τη σημασία που έχουν οι δορυφόροι. Και τέλος το ερευνητικό πρόγραμμα που το αναφέρει η συγκήτρια που πρέπει να συνδυαστεί με όλα τα ερευνητικά εργαλεία. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Ξέρω ότι δεν είναι καινούργια όλα αυτά, αλλά σας πω και εγώ την άποψή μου. Αφού μιλάμε για κλιματολογικές αλλαγές και προσαρμογή αυτές, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ένωση πρέπει να χορηγήσει περισσότερα κονδύλια για τη μείωση των πομπών διοξιδίου παρότι για τα υπόλοιπα. Στη Λευκή Βίβλο της Κομισιόν γίνεται λόγος για τον ορισμό για τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής που έπρεπε να είχε δημιουργηθεί το 2009. Θα ήθελα να γνωρίζω αν δημιουργήθηκε και αν ναι πώς λειτουργεί και αν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κενοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ζαντό. Σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να περιοριστείτε στο δίλεπτο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. Καταρχήν υπογραμμίσω την ποιότητα σχετικές έκθεσεις που έγινε από τον συνάδελφο, από τον συνάδελφο του Επιτροπή Περιβάλλοντος και επίσης ε, και την ποιότητα της έκθεσης της συναδέλφου Ματίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις ε, κατασκευαστικές άδειες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τώρα, τι αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια υποδομή είναι ευάλωτη προφανώς, αλλά και το σύνολο του συστήματος μπορεί να είναι ευάλωτο. Ας φανταστούμε μια χώρα όπως η Γαλλία με πολύ μεγάλη ξηρασία και πραγματικά η Γαλλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υδροελεκτρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τα πυρηνικά. Θα είχαμε λοιπόν μεγάλο πρόβλημα αν είχαμε ξηρασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το θέμα της συμβατότητας κλίματος των ε, υποδομών με την αντίστοιχη συμβατότητα των συστημάτων στις κλιματικ... με τις κλιματικές αλλαγές. Θα μπορούσαμε να έχουμε παρόμοια ανάλυση και για τη Γεωργία. Αυτό εδώ αναφερθήκατε και στο θέμα των μεταφορών, για το θέμα της ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το σύστημα. Δεύτερον, και αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κράτη-μέλη έχουν εθνικά σχέδια προσερμογής και δεν θα πρέπει αυτά να δημοσιοποιούνται. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να συμμετάσχει στο δημόσιο, στην όλη αυτή διαδικασία. Στο πακέτο κλίματος ενέργειας υπήρξε πολιτική δέσμευση ένα τμήμα των εσόδων ε, από τις ποσοστώσεις εμπορίας εκπομπών ε, να ε, χρησιμοποιούνται για το θέμα της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγές. Ίσως λοιπόν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει δέσμευση αυτή και πρέπει να γίνει σεβαστή, να υλοποιηθεί. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στη δέσμευση που ελήφθη στην Κοπενχάγη για την αρρωγή που πρέπει να δίνεται στις χώρες του Νότου. Θα ήταν και αυτό ένα σημαντικό μήνυμα. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σκυλακάκης. Κυλακάκης. Ε, thank Adaptation is inevitable. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσαρμογή είναι κάτι το αναπόφευκτο, διότι οι κλιματολογικές αλλαγές για τα επόμενα 30 χρόνια είναι κάτι που το έχουν προαποφασίσει οι επιστήμονες και άλλοι. Θα χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και στη Λευκή Βίβλο της Κομισιόν δεν προβλέπεται καμία προτεραιότητα Πρέπει όμως απαραίτητος να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα του τι αναμένουμε να συμβεί για να καθορίσουμε προτεραιότητες άλλο τι θα γίνει σε 100 χρόνια και άλλο τι γίνεται ήδη από σήμερα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη. Time frame and for that we need... Χρειάζονται λοιπόν προτεραιότητες και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη έρευνα λόγω της αβεβαιότητας του φαινομένου. Και αυτή η έρευνα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό, ενωσιακό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει σε εθνικό διότι θα γίνουν τεράστιες εξοικονομήσεις κλίμακας όταν γίνεται η έρευνα πανενωσιακός. Αυτό πρέπει να το λέει νομίζω η γνωμοδότησή μας. Τώρα για τα περισσότερα κονδύλια για τον περιορισμό των εκπομπών παρά για την προσαρμογή. Ναι, συμφωνούμε. Τα περισσότερα χρήματα, την τεράστια πλειοψηφία τους δίνουμε για τον περιορισμό και ελάχιστα για την προσαρμογή. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως θα υπάρξουν καθόλου κονδύλια για την προσαρμογή, γιατί μερικοί έχουν την τάση να τα μηδενίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να αναφερθεί στο θέμα. Κανένας? Κανένα. Κομισιόν, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Um, thank you, Mr. Chairman, for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πολύ καλή δουλειά της και που έχει τονίσει ε, κάποια σημαντικά σημεία στους διάφορους τομείς. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η Λευκή Βίβλος ε, εντοπίζει 30 δράσεις που θα υλοποιηθούν στους τέσσερις πυλώνες ε, στην πρώτη φάση. Ενίσχυση της γνωσιακής βάσης, ε, ενίσχυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της των πολιτικών μέσων καθώς και ενίσχυση της ε, διεθνούς συνεργασίας. Για το, τον πρώτο από αυτούς τους τομείς θα μπορούσα να αναφέρω κάποια θέματα που συνδέονται με το κόστος εφαρμογής. Υπάρχουν διάφορα τέτοια προγράμματα, όπως ε, το ΠΕΣΕΤΑ, που εξετάζουν ε, τα, το κόστος προσαρμογής διαφόρων τομέων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει Διάφορε διάφορες έρευνες. Μια έρευνα εξετάζει ιδιαίτερα το κόστος προσαρμογής στον ε, τομέα της έρευνας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία εκτελεί μια στρατηγική που έχει να κάνει με το κόστος προσαρμογής ε, που θα συμπεριληφθεί στις εκθέσεις της. Όσον αφορά την ερώτησή σας για την διευθύνουσα ομάδα, θα ήθελα να σας πω ότι η πρώτη προκαταρκτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περσινής χρονιάς. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας προβλέπεται σε μερικούς μήνες. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις παρατηρήσεις σας. Τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας ε, θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ γρήγορα για να μην ξοδεύω και το χρόνο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια. Νομίζω ότι είναι κατάλληλα και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία δυσκολία να τα συμπεριλάβω. και φυσικά αναμένω και την παρουσίαση των τροπολογιών. Απλώς να αναφερθώ στο κάποια θέματα που είχα να κάνουν με το προήμιο. Αυτά μπορείτε να τα βάλετε ε, στις τροπολογίες. Αναφερθήκατε στις πλημμύρες λόγου χάρη και σε ό,τι αφορά τις γενικές υποδομές. Εδώ αυτή η γνωμοδότηση ζητήθηκε και ε, από την Επιτροπή Γεωργίας ε, να γνωμοδοτήσει αλλά και από την Επιτροπή Μεταφορών. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι ήταν περιορισμένα αυτά που μπορούσα να κάνω εγώ. Πάντως ε, μπορώ να σας πω ότι μας επιβάλλονται κάποια όρια που δεν θέλουμε εμείς να έχουμε αλλά ε, δεν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι παραπάνω και θα ήθελα να το πω αυτό για να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την υποστήριξή της, ε, για την ε, υλοποίηση της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου, 12 η ώρα. Σημείο 25. Γεωργία και αλλαγή του κλίματος. Ο κύριος Όζα Βάγνερ έχει το λόγο. Κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, έστειλε στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου μια σειρά παρατηρήσεων για την, παρουσίαση, για την ε, έκθεση συγγνώμη, του κυρίου Λεφόλ. Είναι καταπληκτική η έκθεσή του γιατί μπορώ να πω ότι με ακρίβεια προσεγγίζει όλα τα θέματα που ε, μας απασχολούν. Και εμείς από τη δική μας Επιτροπή κάναμε τις εξής παρατηρήσεις. Καταρχήν ζητούμε από την Επιτροπή να προβλέψει περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους για την έρευνα και την ανάπτυξη με στόχο να υπάρξουν βελτιώσεις ε, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα στους ε, ακόλουθους ε, τομείς προτεραιότητας. Καταρχήν, παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων, ε, ε, στο μέτρο που το παρουσιάζει και ο κύριος Λεφόλ, δεύτερον παραγωγή και χρήση βιώσιμων λιπασμάτων και αξιοποίηση όλων των γεωργικών αποβλήτων. Αυτά προτείνουμε στον εισηγητή και στη συνέχεια ζητούμε ε, να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν ευρώτερη τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών, γιατί θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επίβλεψη διάφορων φάσεων τη παραγωγή και να βελτιώσουν ε, τη διαχείρισή του με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή σε σχέση με χρήση μέσων που απαιτούνται και ταυτόχρονα να μειωθεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργεια. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις λοιπόν ε, που υποβάλαμε για την πολύ καλή έκθεση του κυρίου Λεφόλ και απλώς πρέπει να προσθέσω κάτι που γνωρίζουν και συνάδελφοι ότι ως τις 2 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών σε αυτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον ε, εισηγητή. Ήθελα να κάνω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις ως ε, σκιώδης συντάκτης νομοδότησης στο θέμα αυτό που συνδέεται άρρηκτα και με την συζήτηση που είχαμε πριν. Ε, είναι προφανές ότι η γεωργία συνδέεται άρρηκτα με τις κλιματικές αλλαγές, με δύο μάλιστα τρόπους. Ε, από τη μια συνδέεται διότι έχει μια σημαντική συμβολή στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ευθύνεται για το 9,3% των συνολικών εκπομπών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη πλευρά έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες ε, συμβολής στους στόχους μετριασμού της, ε, της κλιματικής αλλαγής, με τον περιορισμό βεβαίως αφενός των δικών της εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τις δυνατότητες αποθήκευσης του άνθρακα στο έδαφος και βεβαίως, το είπε και ο εισηγητής πριν, είναι κεφαλαιόδου σημασίας ειδικά για την Επιτροπή μας, με την ε, ενίσχυση της παραγωγής αϊφόρων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ε, ήθελα να σημειώσω βεβαίως ότι πέραν αυτών των επιμέρους στόχων είναι προ, στόχων είναι προφανές και δεν αμφισβητείται από κανέναν ε, ότι ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να ακολουθεί στη γενικότερη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης. Συνεπώς, η πιο, ε, η πιο βιώσιμη προσέγγιση στο θέμα που κουβεντιάζουμε νομίζω ότι πρέπει να στηρίζεται σε μια ε, ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης της ε, περιβαλλοντικής δυναμικής, της περιβαλλοντικής διάστασης της γεωργίας και από την άλλη στη διατήρηση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας ε, του τομέα. Ε, για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία πιστεύω ότι πρέπει να λαμβάνουμε στο σχεδιασμό πολιτικών συνεχώς υπόψη μας το δίπτυχο ε, που ανέφερα και πριν, δηλαδή αφενός των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην γεωργία και αφετέρου των δυνατοτήτων συμβολής στην καταπολέμηση του φαινομένου ως προς το πρώτο, ως προς την επιβάρυνση δηλαδή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στη Γεωργία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλες πιέσεις και προκλήσεις που υφίσταται ο, ο γεωργικός τομέας, ο αγροτικός τομέας, από τον διεθνή ανταγωνισμό, από την φιλελευθερωποίηση των εμπορικών πολιτικών, τη συρρήκνωση του αγροτικού πληθυσμού, ε, και ότι βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, τη χωροταξική κατανομή των κλάδων παραγωγής, τη σταθερότητα της γεωργικής παραγωγής, την ανάπτυξη της δασικής παραγωγής και της ε, ε, δασοκομείας και βεβαίως θα με επιτρέψετε να υπενθυμίσω ως Ευρωβουλευτής από μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου ότι οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται με την ίδια βαρύτητα σε όλη την ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη περισσότερο άμεσες, ορατές και οδυνηρές σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κυρίως στις, ε, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στις χώρες της, της Μεσογείου. ολοκληρώνω με, μία επισήμανση που αφορά, με δύο-τρεις παρατηρήσεις μάλλον που αφορούν στο κομμάτι της συμβολής της γεωργίας στην, στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, μια συζήτηση για τη δυνατότητα επέκτασης του, του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας αερίων στη χρήση γης και στην δασοκομεία. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή και έχοντας κατά έχει επίσης την ανάγκη ταυτόχρονης χρηματοδοτικής στήριξης του τομέα, για να μην τον επιβαρύνουμε ε, περαιτέρω και ασφαλώς το λέει ο εισηγητής μας στη γνωμοδότησή του ε, ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης και παραγωγής χρήσης βιοκαυσίμων, συνδέοντας άμεσα την, τη γεωργία με το κοινοτικό στόχο του 20% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Τίκαου. Να σας θυμίσω να, να προσπαθούμε να περιοριζόμαστε στο δίλεπτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η γεωργία μπορεί πράγματι να έχει, να επηρεάσει, να έχει επιπτώσεις μάλλον να ζημιώνεται από τις κλιματολογικές αλλαγές και επίσης συμβάλλει και στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου αλλά και η ποιότητα των ποσίμων υδάτων σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τα υπόγεια είδα δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τη γεωργία και τις ε, ουσίες που βάλαμε στο χώμα ως λιπάσματα. Πρέπει βέβαια επίσης να αναλύσουμε τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών και επί της ίδιας της γεωργικής παραγωγής. Σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης υπάρχει απερίμωση και στη χώρα μου τη Ρωμανία όλο και περισσότερες μεγαλύτερες επιφάνειες απεριμώνονται. Γι' αυτό έχουν προβλεφθεί με ορισμένα συστήματα άρδευσης ε, στις περιφέρειες αυτές ε, και αυτό θα πρέπει να γίνει η προτεραιότητα της Ευρώπης. Γιατί αλλιώς θα σημειωθεί, θα ξεσπάσει κρίση και για τη διατροφή του πληθυσμού εκεί. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και πρέπει η Επιτροπή μας, που αν δεν με λέγεται Ήτρε, να δώσει στην Επιτροπή Άγκρη Γεώρ στοιχεία που να αφορούν και την τεχνολογία και την έρευνα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιέργειες για χρησιμοποίηση ως βιοκαύσιμα επηρεάζουν γενικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή και εδώ έχουμε μια καλή δρομοδότηση του εξαιρετικού συναντέλφου Στεφάν Λεφόλ. Έκθεση μάλλον. Τώρα για τη δική μας γνωμοδότηση. Πρώτον είναι πολύ θετικό να ζητήσουμε μεγιστοποίηση της χρήσης των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας. Αντίθετα Έχω ορισμένες αμφιβολίες για τις συστάσεις. Γίνεται λόγος για τα βιοκαύσιμα και τα αγροκαύσιμα. Θα έπρεπε η Επιτροπή μας να αποσαφηνίσει ποια είναι τα αγροκαύσιμα επί των οποίων θέλουμε να επιταχυνθεί η έρευνα. Ξέρουμε ότι της πρώτης γενιάς αυτού του είδους τα καύσιμα δεν είναι πολύ αποτελεσματικά και επομένως θα έπρεπε να αποσαφηνίσουμε ποια ακριβώς εννοούμε και ποια θα θέλαμε να τονίσουμε για την έρευνα. Δεύτερον, τα λοιπάσματα, παραγωγή και χρήση των λοιπασμάτων. Ο εισηγητής μίλησε για βιώσιμα λοιπάσματα. Αυτός ο όρος βιώσιμο είναι βέβαια πάντοτε ασαφής. Πρέπει όμως, πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε ότι όλα τα λοιπάσματα που προέρχονται από τη χημειοβιομηχανία πρέπει να περιοριστούν πολύ στη γεωργία ιδίως όταν προέρχονται από υδρογονάνθρακες. Για την έρευνα ζητάμε περισσότερη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων των γεωργών ώστε να γίνεται πιο στοχευμένα. Και τέλος, στα συμπεράσματα της έκθεσης Λεφόλ αναφέρεται ότι η γεωργία εκπέμπει πολύ λίγο διοξίδιο του άνθρακος. Εδώ όμως ίσως θα έπρεπε να διευρύνουμε την έννοια γεωργία και στην ε, βιομηχανία των τροφίμων, διότι όταν ένα γιαούρτι απαιτεί μεταφορά υλικών σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα από την παραγωγή μέχρι την πώληση, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα και αγροτικά επομένως προϊόντα τα οποία μπορεί τελικά λόγω της γενικότερης οικονομίας των τροφίμων που σχετίζεται και με την οργάνωση γενικότερα της γεωργίας να έχουν επιπτώσεις που δεν τις λαμβάνουμε υπόψη ε, με την προηγούμενη έννοια. Θα έπρεπε όλα αυτά να εξεταστούν αν θέλουμε να μειωθεί η εκπομπή αερίων. Ο κύριος Παναγιάτος. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βάκνερ για την εξαιρετική εργασία του. Υποστηρίζω την πρότασή του, δηλαδή να υπάρξει αύξηση των πορών για την παραγωγή των βιοκαυσίμων, όπως επίσης και ότι πρέπει να αγγιθούμε για την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τα οικολογικά πρότυπα και να προσπαθούμε να διατηρούμε μια ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας, της αποδοτικότητας. Νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε στενά και θα είναι επικοδομητική συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στην Κομισιόν στον κύριο Τρίζεν. Κομισιόν, θέλετε το λόγο? Όχι. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνο. Ποιος είναι αρμόδιος για θέματα κλίματος. Όλοι μάλλον. Υπερβολικά πολύ. Α, δεν είναι πρόβλημα κλίματος, είναι πρόβλημα μικροφόνου. Αφήστε να τραγουδήσουν σαν χοροδία, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, το βρήκα το κουμπί. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο συνάδελφος για το προηγούμενο ε, θέμα. Η Κομισιόν ακούει με πολύ ενδιαφέρον αυτά που υπόθηκαν. Φυσικά εργαζόμαστε πάνω σε πολλά από τα ζητήματα που αναφέρατε, διότι είναι ζωτική σημασίας θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν το 2009 εκπώνησε δύο έγγραφα εργασίας για την προσαρμογή στην Γεωργία για να ξεκινήσει η συζήτηση με όλους τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων αυτών από την τροφική λυσίδα. Θα ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή, θα συμμετάσχουμε στην ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της συνέχειας ε, της ε, Λευκής Βίβλου όσον αφορά τη Γεωργία και όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν, η παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων, η αντιμετώπιση των προκλήσεων, το, η αξιολόγηση κινδύνων, το τι θα πρέπει να γίνει όσον αφορά την στήριξη στη γεωργία. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή την επόμενη ΚΑΠ, την επόμενη κοινή γεωργική πολιτική που θα εφαρμοστεί μετά το 2013. Στο μεταξύ, ήδη συμπεριλαμβάνονται στην κοινή γεωργική πολιτική πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη και περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη εποφελούνται από τα μέτρα αυτά. Να αναφέρω ένα παράδειγμα η βιομάζα, η βιοενέργεια πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κάποιοι γεωργοί ήδη λαμβάνουν στήριξη για την παραγωγή βιοαερίου. Η πορεία εδώ είναι πολύ καλή διότι περιορίζουμε τις εκπομπές, βοηθάμε τους γεωργούς να παράγουν ενέργεια και να έχουν έτσι πρόσθετο εισόδημα όταν πολλούν μέρος της ενέργειας που παράγουν. Χρειαζόμαστε όμως χρόνο για να τους εξηγήσουμε για να τους εξηγήσουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται. Αντιμετωπίζουμε και άλλες προκλήσεις. Την παραγωγή τροφίμων σε τιμή που να μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές στην Ένωση ή σε όλο τον κόσμο. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν όλα όσα έχετε να πείτε για την ε, έκθεση του κ. Λεφόρ και θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόζα Βάγνερ, θέλετε το λόγο πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις ε, παρατηρήσεις που ακούστηκαν εδώ και από τους τέσσερις ε, συναδέλφους ε, όσο και με τις διευκρινήσεις της εκπροσώπου της Κομισιόν. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι πολύ στοχευμένες. Νομίζω ότι ουσιαστικά εντάσσονται εδώ στο αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή το σχέδιο γνωμοδότησης του κ. Λεφόλ, αλλά ε, νομίζω ότι είναι και στοχευμένες οι παρατηρήσεις που έρχονται από την πλευρά της Επιτροπής μας. Οι ε, παρατηρήσεις λοιπόν ε, που ακούστηκαν νομίζω ότι θα μας οδηγούσαν στο να διευκρινίσουμε κάποια από τα θέματα που έχω διατυπώσει εδώ στην έκθεση. Έτσι λοιπόν θα σας ευχαριστούσα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου να ε, μπορέσετε να καταθέσετε τροπολογίες έτσι ώστε συγκεκριμένα να μου παρουσιάσετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να συμπεριλάβω στην έκθεση που θα παρουσιάσουμε ως Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλα αυτά είχαμε να πούμε. Λοιπόν, για το ζήτημα, ας περάσουμε το επόμενο σημείο. Ο, ο κύριος Βάγνερ ε, ήδη ανέφερε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 2 Φεβρουαρίου. Το επόμενο θέμα είναι η διακυβέρνηση του ίντερνετ, τα επόμενα βήματα. Πάλι σειρά σας, ε, κύριε Βάγνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι ε, που απασχολώ τόσο πολύ εδώ τους συναδέλφους σήμερα το πρωί. Αλλά πραγματικά ε, μου ανατέθηκε και η εκπόνηση της γνωμοδότησης για τη διακυβέρνηση του ίντερνετ. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέμα, όλα έχουν να το διαδίκτυο. <laughs> περιλαμβάνουν πολλά προβλήματα γιατί πραγματικά το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα ε, και ατομικά και συλλογικά και έτσι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ε, που καλύπτει όρος ίντερνετ διαδίκτυο, όμως εδώ έχουμε να προσεγγίσουμε μόνο το θέμα της διακυβέρνησης του ίντερνετ, δηλαδή ποια είναι η διαχείριση, διακυβέρνηση στο τομέα του διαδικτύου. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί λοιπόν ε, η δική μας γνωμοδότηση. Εγώ ήδη συναντήθηκα με τους συζητητές από τις άλλες ε, πολιτικές ομάδες, συγκεκριμένα με την κυρία Κοχμελίν, την κυρία Τράουτμαν, τον κύριο Φανιστερόι, τον κύριο Λάμπερς και τον κύριο Μπέλετ ε, από την Επιτροπή Πολιτισμού Συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο, ιδιαίτερα καρποφόρος ήταν η συναντησή μας, γιατί εγώ τους παρουσίασα ένα έγγραφο, ένα σχέδιο της έκθεσης και αυτοί μου υπέβαλαν μια σειρά παρατηρήσεων, τις οποίες εγώ φυσικά έχω υπόψη μου τη στιγμή της εκπόνησης. Λοιπόν, για να με μακρηγορήσω και για να ακούσω και τα δικά σας σχόλια, που είναι το πιο σημαντικό, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, το κεντρικό θέμα αυτού του προβλήματος της διακυβέρνησης του ίντερνετ ε, είναι το πρόβλημα ενός ιδρύματος που έχει πολύ συγκεκριμένη ε, νομική υπόσταση, λέγεται ICAN. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που διέπεται από το δίκαιο της Καλιφόρνιας, δηλαδή μιας πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει προνομιακή σχέση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο οργανισμός ε, έχει στα χέρια του ε, την ε, απόδοση των τομέων, των domains και των αριθμών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η φόρμουλα είναι αποδεκτή, αυτό θα συζητήσουμε εμείς. Εγώ να σας πω ότι συμφωνώ με αυτή τη φόρμουλα και με τη διατήρηση αυτού του οργανισμού. Όμως το πρόβλημα έγινε στη δομή αυτού του οργανισμού και τις ξεχωριστές σχέσεις που έχει με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και αναθεωρήθηκε πρόσφατα μέσω μιας σύμβασης που υπεγράφει πρόσφατα. Δηλαδή, το πρόβλημα έγκυται στο να ανοίξει αυτός ο οργανισμός που έχει στα χέρια του κάτι πολύ σημαντικό όπως το θέμα της ε, ε, απονομής τομέων και νούμερων στον κόσμο. Μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό, ένα αγαθό δημόσιο χαρακτήρα που αφορά την ανθρωπότητα στο σύνολό της και που παρόλα αυτά τη διαχείριση την έχει αναλάβει ένας μόνο οργανισμός που επιπρόσθετα είναι και ιδιωτικό και ελέγχεται από την κυβέρνηση ενός μονοκράτους των ΗΠΑ. Εμείς εδώ ως ε, μέλη των Ευρωπαϊκών Οργανισμών πρέπει να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε έναν τρόπο έτσι ώστε αυτή η διαχείριση του ICAN να είναι πιο πλουραλιστική και πιο ανοιχτή. Αυτό είναι το κύριο θέμα ε, και ο στόχος της παρέμβασής μας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ποιο είναι κατάλληλοι τρόποι και φυσικά εγώ προς αυτή την κατεύθυνση εκπονώ την ε, έκθεσή μου, αλλά αν έχετε οποιασδήποτε προτάσεις ε, θα σας ευχαριστούσα. Επιμένω να αναζητήσουμε με ποιο τρόπο η Ευρώπη θα είναι περισσότερο παρούσα, με πιο προσδιορισμένο τρόπο, στην διακυβέρνηση αυτού του συλλογικού αγαθού. Και βέβαια θέλουμε να ενισχύσουμε και τους πολυμερείς ελέγχους επί του οργανισμού αυτού, ο οποίος είναι τόσο ιδιαίτερος ε, και έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, όπως σας είπα. Από την άλλη μου φαίνεται πολύ σημαντικό να προσεγγίσουμε το θέμα του λεγόμενου φόρουμ της κυβέρνηση του διαδικτύου. Αυτό το φόρουμ, το οποίο τελευταία συνεδρία έλαβε χώρα σε μία πόλη της Αιγύπτου, πέρσι τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί. Είναι πολύ σημαντικό ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, να στοιχηματίσουμε περ αυτού του φόρουμ διακυβέρνηση του διαδικτύου. Γιατί, γιατί το διαδίκτυο στην προσωπική και συλλογική μας ζωή, όπως σας είπα, ε, υπάρχει και αποτελεί ένα τόπο όπου συγκεντρώνονται μεγάλα και δημόσια αλλά και ιδιωτικά συμφέροντα. Και αυτό το φόρουμ διακυβέρνηση του ίντερνετ τελικά έχει ως ε, σκόπο να ε, διαχειρίζεται όλα αυτά τα συμφέροντα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το μεγάλο φόρουμ. Ε, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ίντερνετ, δεν μπορούμε να το ξημειώσουμε με κανένα άλλο μεγάλο θεσμό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο και αυτό το φόρουμ διακυβέρνησης του ίντερνετ, όπως σας είπα, έχει ως στόχο να εκπροσωπεί όλα τα συμφέροντα. Υπάρχει ένα ε, πολύ καλό σύστημα συζήτησης για την προσέγγιση των προβλημάτων. Όπως ε, μας είπε και η κυρία Τράουτμαν ε, στην έκθεσή της, μας παρουσίασε στην προηγούμενη συνάντηση Επιτροπή Ήτρα, αυτό το φόρουμ θα συναντηθεί και πάλι περί τα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο στη Λιθουανία. Είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα να έχουν καθορίσει ποια θέση θα ακολουθήσουν ε, για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και ε, έχοντας τη θέση αυτή να συμμετάσχουν σε αυτό το πολύ σημαντικό ραντεβού. Βεβαίω ε, και είμαι ανοιχτό να ακούσω τις ε, παρατηρήσεις και τις ε, προτάσεις σας και ήδη να σα πω ότι 17 Μαρτίου θα έχουμε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων και θα ήθελα να ζητήσω από τους φίλους και συναδέλφους να μου δώσουν ονόματα αν ενδιαφέρονται προκειμένου να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τράουτμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγνερ και το σύνολο των συναδέλφων που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Και εγώ ως καλής ε, βρίσκομαι στο πλευρό του για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Σκιώδη συγγήτρια, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του χρονοδιαγράμματος και θα έχουμε στο Βίλνιους ε, και πάλι τη συνάντηση του φόρουμ. Ε, το πρώτο, η πρώτη συνάντηση του φόρουμ έγινε στην Αθήνα και εκεί δηλώσαμε την πρόθεσή μας ε, το διαδίκτυο να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους, να έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση και φυσικά στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών. Στο Βίλνιους ε, και το συστήσαμε αυτό το θέμα χθες σε άτυπη συνάντηση όπου περιβρίσκονταν ε, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της Ισπανικής Προεδρίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήσαμε λοιπόν για το πώς προχωρούν οι προετοιμασίες ε, της ε, Επιτροπής Εργασιών ε, για το Φόρουμ και αναφερθήκαμε στις μελλοντικές συναντήσεις. 29 και 30 Απριλίου θα λάβει η χώρα μία συνεδρίαση του Eurodic της πλατφόρμας όπως συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές, τα εθνικά IGF, το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και άτομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο στη Μαδρίτη. Η συνάντηση αυτή θα υποστηριχθεί από την Ισπανική Προεδρία. Αλλά οι συνάδελφοι από την Ισπανία μας είπαν ότι Τη η Ισπανία ακόμη δεν έχει καθορίσει σε ποιο βαθμό θα τεθεί ε, ως προτεραιότητα το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Όμως εμείς θα θέλαμε το Βελνίους να είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη συνέχιση του φόρουμ, ε, για ε, την μεταρρύθμιση του οργανισμού ICAN και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που η Ισπανική, η Προεδρία να μπορεί να θέσει ψηλά στην μερική διάταξή της. Αυτό είναι σημαντικό για το σύνολο των χωρών της διεύρυνσης και είναι σημαντικό για το τι θα πούμε στις αφρικανικές χώρες. Ως ε, συνέχεια των ανταλλαγών που είχε η αντιπροσωπεία μας ε, στο IGF, e ε, στο φόρουμ, Θέλουμε να προετοιμάσουμε για το Vilnius ε, ένα workshop ε, όπου θα συμμετάσχουν ε, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων από τις Αφρικανικές χώρες. Και καθώς συναντηθήκαμε με μια αντιπροσωπεία από τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής και συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους από τη Βραζιλία και την Ινδία που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε τα θέματα αυτά για την προετοιμασία. και στις 9 Φεβρουαρίου θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να συνοδεύσει την Επιτροπή στην προπαρασκευαστική συνάντηση για το Βίλνιους και κατόπιν τον Ιούνιο έχουμε προπαρασκευαστική συνάντηση με τους εκπροσώπους ε, των κοινοβουλίων προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτό το workshop στο ε, IGF στο Βίλνιους 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, όσο λοιπόν δρομολογείται η έκθεση και ε, εμείς ε, με την Ισπανική αλλά και με τη Βελγική Προεδρία ε, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες ε, θα έχουμε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν και να διευρύνουμε και την επιρροή μας. Για να κλείσω, Πρόεδρε, εμείς ε, θεωρούμε ότι το διαδίκτυο είναι δικαίωμα η πρόσβαση στο διαδίκτυο και έτσι λοιπόν και από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, αλλά και εμείς εκφράζουμε κάποιες ανησυχίες ε, νομικού χαρακτήρα, όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, η ασφαλής πρόσβαση και ε, επί της σύμβασης για τον έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αυτά είναι σημαντικά από ευρωπαϊκή σκοπιάς αν μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα. Έχουμε ε, κάποιες ακόμα παρεμβάσεις. Ο συνάδελφος Νίστελ Ρόι, παρακαλώ να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο εισηγητής ε, και να περιοριστούμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ίντερνετ. Ε, είναι ε, μεγάλο το έργο αυτό. Η ενημέρωση δηλαδή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας σχετικά με τον τομέα αυτών. Μπορεί να υπάρχουν δέκα ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο που να ξέρουν περί τίνος πρόκειται, μάλλον όχι περισσότεροι. Και αναφέρθηκε ήδη αυτό στην ε, πρόταση λοιπόν αυτή που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. Τίθεται το θέμα της αρμοδιότητας ε, και είναι πολύ καλό ότι αναφέρονται τα θέματα αυτά. Και θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να συμμετάσχουν στις ενέργειες αυτές. αναρωτιόμαστε εάν το φόρουμ για τη διαχείριση του ίντερνετ που δεν είναι ε, νομικά δεσμευτικός φορέας, εάν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Βρίσκω ότι είναι πολύ ωραίο το Κοινοβούλιο, έχει λέγει, αλλά θα πρέπει να καταλάβει το Κοινοβούλιο ότι συζητάμε το θέμα αυτό και θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι για, μια σειρά μέτρων ε, θα επιλέξουμε να προχωρήσουμε, ενώ άλλα, με άλλα δεν θα ασχοληθούμε. Μετά την Κοπεχάγη υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις ε, ιδέες μας με, δεσμευτικές, ε, δεσμευτικά μέσα. Είδαμε τι έγινε με την Κομεχάγη, σκεφτόμαστε με επιστημονικό τρόπο, αλλά η Κίνα ε, ερμηνεύει αλλιώ τις αρχές, ερμηνεύει αλλιώς τα πράγματα και απέχει πολύ από τις αρχές μας. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά το διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε σε συγκεκριμένα θέματα και θα πρέπει μαζί με την ICAN, ε, ε, την ομάδα εργασίας ε, που ασχολείται με την ατζέντα του φόρουμ, θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους αυτούς, να δούμε πού θα οδηγηθούμε και... Αν αναθέσουμε σε κυβερνητικό επίπεδο μια σειρά θεμάτων και τελικά δεν γίνει τίποτα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το πακέτο του διαδικτύου καλύτερα μέσω του, της ICAN. Και άλλωστε δεν χρειάζεται να ξαναρχίσουμε εκ νέου τη συζήτηση. Όσον αφορά αυτά που είπε ο εισηγητής, βρίσκω ότι πολύ σωστά συνόψε τις θέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω δύο λόγια για τη δυνατότητα ανοίγματο στο ICAN. Γνωρίζετε ότι πριν κάποιους μήνες γίναμε μάρτυρες μιας θετικής εξέλιξης το έκανα δεν ε, έχει ε, κλειστή σχέση με την ε, κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις σας ότι πρέπει να διασφαλίσουμε αυτό το δημόσιο αγαθό που είναι το διαδίκτυο, όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενεργή, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος να ε, δημιουργήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη του διαδικτύου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα λαμβάνει η χώρα μια διαδικασία για ε, το να χρησιμοποιούνται τα διάφορα αλφάβητα, το κυριλικό κτλ. Έτσι λοιπόν, καθώς μιλάμε για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα που να είναι αρκετά ευέλικτη για να μην ε, προκαλέσουμε μπλοκή στη διαχείριση αυτού του αγαθού. Κυρία Τικάου. Δεν ε, θα ήθελα να μακρηγορήσω. Επιτρέψτε μου να αναφέρω το ότι εδώ πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τώρα τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας που δίνει επιπρόσθετες ε, αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συζήτηση που έλαβε η χώρα τους τελευταίους μήνες ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των χρηστών. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ελευθερία στο διαδίκτυο. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει επικοδομητικά σε όλη αυτή τη συζήτηση. Από εκ μέρους της ε, Μελλοντικής Επιτρόπου αναμένουμε εμπλοκή σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι μέλος μιας επιτροπής που θα ήθελε να συμμετέχει σε όλα αυτά τα φόρουμ και τις ε, συνεδριάσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν συγχαίρω τον συγητή και φυσικά να του πω ότι έχει την υποστήριξή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη παρέμβαση από την Κομισιόν, ο κύριος Νίμπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Η ανάλυση για την ICAN, ε, ναι, πρόκειται για ιδιωτικό φορέα και ναι, διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό. Στη δήλωση δέσμευσης ανάμεσα στη ε, κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ΆΙΚΑΝ είδαμε ότι για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ε, κάνει ε, ένα πρώτο άνοιγμα, αλλά εκ των υστέρων θα αποδειχθεί πώς θα λειτουργήσει αυτό. και δεν είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει μόνο τους, ε, την πλευρά της ICAN. Αυτό είναι η μία σημαντική παρατήρηση. Η δεύτερη είναι το IGF. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στηρίζουν απόλυτα τη συνέχιση του IGF, του ε, Φόρουμ για τη Διαχείριση του ε, Διαδικτύου, ε, μπορούμε να καλύψουμε πληθώρα θεμάτων και είμαστε ευγνώμενες που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή και που έχει δώσει πολύ περισσότερη αξιοπιστία στην Κομισιόν ότι η ευρωπαϊκή παρουσία ήταν ισχυρή και αποτέλεσε σημεία αναφοράς για τη συμμετοχή βουλευτών από τις κυβερνήσεις άνω κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είδα τον κύριο Τουσνόφσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας είναι πολύ δύσκολο αυτό που ακούσαμε. Το περιεχόμενο βέβαια είναι τέτοια φύση που είναι δυσνόητο, αλλά χαίρομαι γιατί η συζήτηση υπήρξε ανοιχτή και πρέπει να συνεχιστεί έτσι ελεύθερα. Πρέπει όμως να γίνει και μια θεσμοποίηση του τεράστιου αυτού φαινομένου. Όπως είπε και ο κύριος Βανίστελ Ρόι, κανείς σχεδόν δεν καταλαβαίνει περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πριν από 10 χρόνια όταν πρώτο ενδιαφερθήκαμε για το ίντερνετ, ε, κυρίως πανεπιστημιακοί ασχολούνταν με αυτό. Τώρα όμως έχει πάρει άλλες διαστάσεις και πρέπει να υπάρξει κάποια διευθέτηση, πρέπει να το συζητήσουμε, να μιλήσουμε, αλλά δεν ξέρω με τι ακριβώς τρόπο. Καλό είναι βέβαια η Ευρώπη να έχει κάποια άποψη και να προασπίσει τα συμφέροντά της, αλλά δεν πρέπει να παρέμβει για όλα, δεν μπορεί εξάλλου. Για να μην παραμείνει το θέμα δέσμιο μόνο της θεσμικής πλευράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θέρμα. Κύριε Σόζα Βάγνερ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Να πω στην κυρία Κάπμαν ότι φυσικά θα στην Ισπανία θα προβώ τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μάθω α, ουσιαστικά σε ποιο επίπεδο θα λάβει χώρα η συνάντηση στη Μαδρίτη, ποιοι θα συμμετάσχουν και επίσης πέρα από μια συμβουλή λαμβάνω μια οδηγία από σας εδώ να δείξουμε σοφροσύνη, να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή είναι η οδηγία που λαμβάνω εδώ από σας και θα προσπαθήσω να την αντικατοπτρίσω και στην εκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας εύχομαι. Καλό διάλειμμα για το γεύμα. Και θα τα